Dear uh, Vice Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εθνικοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι ως Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής. Σε αυτό το Ευρωφόρουμ το 2015. Αυτό το φόρουμ είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε με το τρίτο τμήμα ε, διαμόρφωσης πολιτικής και με ε, την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Πολιτικών που το κάνουμε κάθε χρόνο με πανεπιστημιακούς, με την ελληνικά κοινοβούλια για να ανταλλάξουμε απόψεις να αφορά τις εξελίξεις ε, σε θέματα αστικού δικαίου και δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Έχουμε 13 εθνικούς βουλευτέ εδώ σήμερα τους συγχαίρω που επέδειξαν ενδιαφέρον για ένα τέτοιο σημαντικό κλάδο του δικαίου. Συνέπεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Πολλά και περισσότεροι Ευρωπαίοι περνούν τα σύνορα. Εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος, παντρεύονται κάποιον πολίτη άλλου κράτους μέλους ή απλά ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος. Υπάρχουν βεβαίω ε, και συνέπειε σε επίπεδο ποινικού δικαίου από αυτή την κινητοποίηση, ε, από αυτή την κινητικότητα μάλλον. Αλλά από την άλλη μεριά πολλές φορές το ότι πολλές φορές ε, αυτοί οι μεταγενόμενοι πολίτες έρχονται σε επαφή και με τις ρυθμίσεις του αστικού δικαίου, χωρίς από το ποινικό δίκαιο. Και ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει με τα ποινικά δικαστήρια. Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κληρονομούν, οι παντρεύονται, ή απλώ εργάζονται σε κάποια άλλη χώρα έρχονται σε επαφή με τις αστικές ρυθμίσεις του άλλου κράτους μέλους. Η ΔΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα επαρκές πλαίσιο και να υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ των ρυθμίσεων του ενός κράτους και του άλλου. πούμε, το είπαμε ότι ήταν μια ρύθμιση που έπρεπε να γίνει και επίσης και άλλη ρύθμιση ε, για τους πολίτες που έχουν ε, ιδιοκτησία σε περισσότερα κράτη-μέλη και έτσι τελικά να ρυθμίζεται καλύτερα η υπόθεση της κληρονομικής διαδοχής τους με τίποτα δεν είναι τα πράγματα τέλεια γιατί ακόμα σοβούν πολλά προβλήματα Περίπου όσον αφορά κάποιες διοικητικές ε, διαδικασίες για αυτούς τους ε, ε, διακινούμενους Ευρωπαίους και επομένως αυτό που θέλουμε σήμερα να πετύχουμε είναι να δούμε τι έχουμε πετύχει, τι προβλήματα έχουμε, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ και όλους όλους με τηλεσυνεδρίαση παρακολουθούν την ε, συνεδρίασή μας. Περιμένω πως και να ακούσω ότι έχουν να πούνε οι πυρογνώμονές μας. Τώρα, ο αντιπρόεδρός μας θα λάβει τον ε, λόγο. Είναι ο αντιπρόεδρος μας που έχει την ε, ευθύνη των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια ο κύριος Μπάλκαρθελ. Και καλώς ορίσατε και, κυρία Ντελό Εσείς κύριε Μπάλκαρθελ τώρα το Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι για μένα είναι μεγάλη μου χαρά το να ξεκινώ αυτό το φόρουμ που αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες που θα κάνει με τις προσπαθειές μας στη ζωή των Ευρωπαίων πιο εύκολη να συσφίξουμε και τις σχέσεις με τα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια. Όπως είπε ο πρόεδρος Σβόποντα, έχουμε 13 συναδέλφους από τα εθνικά κοινοβούλια. Καλώς όρισαν λοιπόν ε, οι συναδέλφοι από αυτά τα 19 εθνικά κοινοβούλια. Βέλγιο, Κύπρος, Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετωνία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβανία, Ισπανία και Σουηδία. Και επαναλαμβάνω, καλώ όρισαν. Επίσης έχουμε εδώ οκτώ προέδρους και αντιπροέδρους κοινοβουλευτικών νομικών επιτροπών. Θεωρώ πάρα πολύ θετικό το ότι μπορούμε τώρα να μιλήσουμε στους του των Κοινοβουλίων, γιατί το θέμα μας, το σημερινό βρίσκεται στην καρδιά των σχέσεων, των σχέσεων διακυβέρνησης στην ε, Ένωση. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σήμερα είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες όσον αφορά την δικαστική συνεργασία, όσον αφορά διάφορα θέματα διασυνοριακά και αυτό από τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Οπότε ε, προκειτού για θέμα κοινή αρμοδιότητα, δηλαδή Ευρωπαϊκή και Εθνική. Άρα, ο όγκος της κοινοτικής νομοθεσία, όσον αφορά το ιδιωτικό διεθνέ δίκαιο σήμερα είναι αρκετά εκτεταμένο. Πάντως, περισσότερες από αυτές τι αρμοδιότητε. ακόμη βρίσκονται σε επίπεδο εθνικής δικαιοδοσίας. Η ΔΕ Ένωση με την εναρμόνιση των νόμων και νομοθεσιών μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, είναι σημαντικό να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου για τη διακίνηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών. Και έτσι θέλουμε να δούμε το πώς θα έχουμε όλο ένα και πιο πλήρες διασυνοριακές σχέσεις. Δηλαδή να φτιάξουμε γέφυρες μεταξύ των διαφορετικών ενόμων τάξεων. Και ξαναλέω, κατασκευή γεφυρών. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εθνικές παραδόσεις. Έτσι θα πρέπει να δούμε πώ θα συντεριάξουμε τα πράγματα. φέτο, δε έχουμε όπως και ε, άλλες χρονιές αυτές τις δύο ετήσιε συναντήσει. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δηλαδή ό,τι προκύπτει από τις δράσεις των ε, φυσικών προσώπων, από όσα κάνουν διακινούμενοι ε, και διαβαίνοντας κάποια σύνορα. Μιλούμε για όλους τους κλάδους του αστικού δικαίου. Ό,τι προκύπτει από τις ε, σχέσεις και πράξεις των προσώπων. Παραμένει το αστικό δίκαιο, εθνικό δίκαιο. Κάθε χώρα, κάθε κράτος μέλος έχει τους νόμους του που προβλέπουν το πώς θα επιληθεί οποιαδήποτε διαφορά. αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κάποια σύγκρουση αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεων στο μέλλον Πάντως, συνήθως οι συνήγοροι προσφεύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που πρέπει να λύσουν. Και τότε, ανάλογα με το εφαρμοστείο δίκαιο, προσπαθούν να πετύχουν την πιο ευμενή τους ε, απόφαση. Αυτό λέγεται forum shopping. Το θέμα είναι τώρα, η ερώτηση για τη σημερινή μα συζήτηση, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των Ευρωπαίων. Σε κάθε περίπτωση που έχουμε διάφορες υποθέσεις ή διαφορές διασυνοριακές. Οπότε, η διαφορες διασυνοριακε αρχή, η πηξίδα μας εδώ, είναι η αρχή τη επικουρικότητα. Όπως ξέρετε, εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών 2012-2014 και στην Επιτροπή των Περιφερειών εκεί έμαθα καλά την αρχή της επικουρικότητας. Ήμασταν κατά κάποιο τρόπο εμείς οι φύλακες της αρχής της επικουρικότητας. Οπότε προσπάθησα να δω πώς θα υπάρχει δημοκρατικός ένωσης από το κοινωτικό δίκαιο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί τις αρμοδιότητές της και τα θεσμικά όργανα να είναι αποτελεσματικά και πάντοτε να δρουν εποφελία των Ευρωπαίων πολιτών. Για να δούμε τώρα τι πάνε να πει επικουρικότητα. Πρώτα πρώτα, η επικουρικότητα βάζει όρια στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αντίθετα η επικουρικότητα όταν υπάρχει προσθέμενη αξία θα πρέπει να προκαλεί ευρωπαϊκή δράση σε ε, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Και τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω τέτοιες αρμοδιότητες, οπότε εγώ θα συνεχίσω το έργο μου. Και Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ πρόεδρε, είμαστε πεπισμένοι ότι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επίπεδων διακυβέρνηση αλλά και των επιμέρου θεσμικών οργάνων πρόκειται να μας ε, οδηγήσει στην ε, πιο άρτια νομοθεσία. Και στο φόρουμ εδώ, στη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια, έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Επίσης, είμαι πεπισμένος ότι δικαιολογείται πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ασχοληθεί με το αστικό δίκαιο. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις συναρμοδιότητες, αλλά πάντοτε πρέπει να προχωρούμε με μεγάλη προσοχή και σε τακτά διαστήματα να ε, αναθεωρούμε το τι έχουμε κάνει. Μα δεν είναι τυχαίο ότι για το αστικό δίκαιο έχουν διαβαστεί στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερε αρμοδιότητε από ό,τι σε άλλου κλάδου του δικαίου και αυτό αφορά επίσης και το οικογενειακό δίκαιο. Το οικογενειακό δίκαιο είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Το τι γίνεται στην πράξη σε κάθε κράτος μέλος. Ε, δεν είναι στεγανή η κατάσταση. Υπάρχει επιρροή και από το εξωτερικό. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιορυθμίες και οι ιδιοτυπίες κάθε κοινωνίας που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές σεβαστές και σε ένα τέτοιο σημαντικό τομέα όπως το δίκαιο. Γι' αυτό μιλώ για τις γέφυρες μεταξύ των ενόμων τάξεων. Πέραν της ε, εναρμόνισης που είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα αναγνωρίζει η συνθήκη. Γι' αυτό και απονέμει στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα του να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε ένα εξάμεινο από όταν περάσει ε, κάποιο νομοθέτημα σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, στο άρθρο 3, σε σχέση με την ε, δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, η Συνδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 81, ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναπτύξει δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις ε, όσον αφορά τις διασυνορικές υποθέσεις. καλύπτει σε όλο το αστικό δίκαιο, το άρθρο 81 αυτής της συνδίκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επίσης ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόκειται ε, με την συνήθεια νομοθετική διαδικασία να προβούν σε λήψη μέτρων φερειπίν σε αμοιβαία αναγνώριση ε, για τις ε, δικαστικές αποφάσεις ή άλλου είδους αποφάσεις ε, ή για διαβίβαση ε, εγγράφων δικογραφίας ή άλλων νομικών εγγράφων, συνεργασία, ε, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, άρση κάποιων φραγμών για την εύρεθμη λειτουργία της πολιτικής δικονομίας και σε άλλα θέματα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτά όσον αφορά το αστικό δίκαιο για τις ε, υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Και έτσι να είναι πιο εύκολη η ζωή των Ευρωπαίων. Τώρα θα ε, δούμε πώς είναι δυνατόν σε, σε τρία τμήματα να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πηγάζουν από το άρθρο 81. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάντως, κάθε νομοθετική πράξη είναι τμήμα των εγγράφων που υποχρεωτικά θα πρέπει να διαβιβάζονται στα Εθνικά Κοινοβουλία. Αυτό ορίζεται από το άρθρο 12 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση όσον αφορά τις αποφάσεις για κάποια ζητήματα οικογενειακού δικαίου που έχουν συνέπειες διασυνοριακές. Εν κατακλείδη, παρακαλώ να ακούσετε το εξής. Με συνήθεια νομοθετική διαδικασία λαμβάνονται αυτά τα μέτρα και εάν δεν έχουμε ένσταση από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε δε ότι τελικά η κυβέρνηση, η διοίκηση η εθνική και η περιφερειακή θα υλοποιήσει και θα εφαρμόσει την κοινωνική νομοθεσία. Γιατί οι εθνικέ αρχές και οι δικαστικές είναι πιο κοντά στον Ευρωπαίο. Εκείνοι επομένω θα δουν ποια είναι η κατάλληλη λύση σε περίπτωση ενδική διαφοράς, ακόμα και αν πρόκειται για διασυνοριακή υπόθεση. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ευρωβουλευτέ, αλλά και οι εθνικοί βουλευτές να συνεργάζονται για τα θέματα της νομοθεσίας. Όλα αυτά είχαμε κατά νου όταν ε, διοργανώσαμε αυτήν την ε, συνάντηση με την ε, νομική μας επιτροπή σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και έχουμε κάποιους πανεπιστημιακούς, κάποιους επαγγελματίες του δικαίου, κάποιους εμπειρογνώμονες τελικά, οι οποίοι μπορούν με τα λόγω γνώσεως να μας εξηγήσουν όλα αυτά τα οποία ε, χρειαζόμαστε να ακούσουμε να, και πρέπει να συζητηθούν αυτά μεταξύ Ευρωβουλευτών και Εθνικών Βουλευτών ούτω ώστε στο μέλλον η νομοθετική διαδικασία να είναι πιο πλούσια, πιο αποδοτική και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Και πριν καν αρχίσουμε εγώ σας συγχαίρω γιατί θεωρώ ότι είναι εγγυημένη επιτυχία από την παρουσία σας εδώ. Και βέβαια τελειώνοντας την εισήγησή μου να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς που βοήθησαν να διαβεβαιωθούν τα όσα είπα εγώ. Πρόεδρος, Σβόμποντα. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ίνες Ερμίνια Αγκινέρα από πλευράς της Λετωνικής Προεδρίας. Εκπροσωπεί το Συμβούλιο. Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Αξιότιμοι συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μου δίνετε η ευκαιρία να σας παρουσιάσω το θεματολόγιο της Λεπτονικής Προεδρίας σε θέματα αστικού δικαίου. Έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους στο νέο Κοινοβούλιο και η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε η πρόκληση για μας είναι να ε, κινήσουμε τη διαδικασία ενός ε, νομοθετικού κύκλου από πλευράς ε, του Συμβουλίου. Η ευχανόμενη ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά αναπόφευκτα μας οδηγεί σε αυξανόμενο αριθμό διασυνοριακών υποθέσεων, οπότε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και το εταιρικό δίκαιο είναι πολύ σημαντικά ζητήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκαιο είναι ένας ε, τομέας ε, που συνδέεται λένε και περισσότερο με την ε, οικονομία αλλά και με την ανάπτυξη και ενίσχυση της διεθνούς αγοράς. Γι' αυτό η πρόθεση της ανάπτυξης έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα για την Προεδρία μας. Προαγάγουμε λοιπόν και το θέμα της ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για διάφορα βασικά νομοθετήματα στον τομέα του αστικού ε, και του εταιρικού δικαίου. Θα ήθελα να να αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα. Ε, ο κανονισμός για τα δημόσια έγγραφα είναι ύψιστη προτεραιότητα για μας θα πρέπει οι Ευρωπαίοι νομοθέτε να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο ώστε να μειώσουν την γραφειοκρατία και να διευκολύνουν ε, την ελεύθερη κυκλοφορία. Ένα απλοποιημένο μητρό για τα δημόσια έγγραφα θα είναι μια σημαντική συμβολή και ένα σημαντικότατο βήμα προ τα μπρο. Οι συζητήσει ε, για τα δημόσια έγγραφα, για τον κανονισμό αυτό δηλαδή, υπήρξαν περίπλοκέ ε, μέχρι στιγμή, μέχρι τα τέλη του 2014. Κατάφεραν να συμφωνήσουν οι Υπουργοί Δικαιοσύνη για μια ε, προσεκτική προσέγγιση, να μειώσουν δηλαδή το πεδίο εφαρμογής ε, του κανονισμού στα δημόσια έγγραφα. Στην πράξη βεβαίως μπορεί να αποδειχθεί ότι εξυπηρετεί τους στόχους του το κανονισμός, ότι διευκολύνει τη ζωή των πολιτών και στη συνέχεια ε, παραμένει ανοιχτό φυσικά το ζήτημα της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ συζητήσει στο Συμβούλιο είναι το θέμα της εξωτερικής αρμοδιότητας, ε, κυρίως ε, υπό το φως της πρόσφατης απόφασης 1.13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πέντε ομάδες εργασίας ε, καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Ο στόχος είναι μια μερική συμφωνία για το κείμενο στις 13 Μαρτίου ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη. Είναι εντατική δουλειά ε, στο Συμβούλιο για να εκπληρωθεί αυτό ο στόχο. Επιπροσθέτω, είμαστε πεπισμένοι ότι θα καταλήξουμε συμφωνία Βουλευτική Προεδρία τον Ιούνιο Ανοίγοντα έτσι και μια νέα δυνατότητα ε, εκείνης των διαπραγματεύσεων για αυτό το θέμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια άλλη προτεραιότητα για τη δική μας Προεδρία είναι αναθεώρηση του κανονισμού σε σχέση ε, με την ε, εγκαθίδρυση διαδικασίας για τη ρύθμιση μικρών, μικρόποσων αξιώσεων αυτό που επιδιώκουμε είναι να λάβουμε υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Ε, στα τέλη του 2014 συμφωνήσαμε σε μια θέση του Συμβουλίου και είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε μέχρι το τέλος της Προεδρίας να καταλήξουμε σε συμφωνία. Επίσης, έχει προγραμματιστεί επίσημα να εγκριθεί ο κανονισμός για την αφαιρεγγιότητα. Επίσης στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης ε, το Μάρτιο είμαστε ε, ε, ικανοποιημένοι διότι για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφαιρεγγιότητας θα έχουμε σύντομα ένα σύστημα που να προσαρμόζεται στις ανάγκες της οικονομίας και έτσι θα συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα βελτιώσουμε την ικανότητα της εσωτερική αγοράς να αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Οι συνομοθέτες θεωρούν ότι το παρά το κανονισμός της αφαιρεγγιότητας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αγαστής συνεργασίας και δείχνει καταδεικνύει την ικανότητά μας να βρίσκουμε ικανοποιητικέ λύσεις για να τονώσουμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την δυνατότητα επίσης θέσπισης ενός κοινού δικαίου πολίσεων. Μέχρι τούδε δεν έχουν τελεσφορήσει οι προσπάθειές μας όμως και μετά την απόσυρση της πρότασης για το δίκαιο πολίσεων ε, στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015 έχει προανακοινώσει ε, την κατάθεση πρότασης για το ψηφιακό περιεχόμενο ανταυτού. Ε, στα, στη Ρήγα τον Ιανουάριο του το 2015 έγινε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων. Ο πρόεδρος Σφόποντα αναφέρθηκε σε μια πιθανή λύση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου, διότι ένα τέτοιο νομοθέτημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα διευκόλυνε τη ζωή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ε, σε σχέση τώρα με, τη σχέση, με την δικαιοσύνη, σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, θα ήθελα να επιμείνω ε, στις προσπάθειες που κάνουμε για να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ε, αυτό νομίζουμε είναι σημαντική συμβολή στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ εν συντομία στα ζητήματα οικογενειακού δικαίου που εντάσσονται στην ίδια στις προσπάθειές μας, ε, παρότι αποτελούν ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν ότι κάνουμε σημαντικότατες προσπάθειες, ούτως ώστε ταχύτατα να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, για την προσχώρηση της Σύμβασης της Χάγης για την απαγωγή των παιδιών από πλευράς 8 τρίτων χωρών. Ε, συζητούνται όλα αυτά τα ζητήματα στο Συμβούλιο, αλλά υπάρχει και ένα νέο κύμα ε, διαπραγματεύσεων για τη γονική ευθύνη, για τα ζητήματα γαμικών καθεστώτων, για τα διασυνοριακά διαζύγια. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφότου εκπνεύσει η περίοδος προβληματισμού πολυβράς των κρατών μελών. Για το εταιρικό δίκαιο διαπιστώνουμε ότι έχουμε την νομοθεσία σε σχέση με τα δικαιώματα των μετόχων και την ενιαία Ευρωπαϊκή Εταιρεία και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Θα ήθελα εν κατακλείδη να τονίσω ότι τα ζητήματα ιδιωτικού διεθνού δικαίου έχουν ιδιαίτερη σημασία για κάθε έναν πολιτή, διότι επηρεάζουν ε, και την ιδιωτική μα ζωή αλλά και τη δουλειά μα σε καθημερινή βάση και ω εκ τούτου θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε ευρωπαϊκέ και ε, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ε, ε, να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία για τους πολίτες ε, και να υπάρχει ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία για τις οικογένειες και για ζητήματα που σχετίζονται με τα παιδιά. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και ελπίζω το σημερινό εργαστήρι θα μας φέρει ένα, ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση αυτών των στόχων. Thank you, for, for your... Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου για τα καλά σας λόγια, για τα γενικά σας λόγια και τώρα να κοιτάξουμε το πρώτο τμήμα της σημερινής συνεδρίας, της λιγότερη γραφειοκρατία για τους μετακινούμενους πολίτες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον ε, καθηγητή προσε... Ε, Φανχάιν από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ να μας κάνει την εισαγωγή σε 10 λεπτά, αν γίνεται. Έχετε το λόγο λοιπόν. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές. Να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω την δυνατότητα να σας παρουσιάσω μία μελέτη την οποία και έχω καταρτήσει με την Γκίζελα Ρουλ από το Πανεπιστήμιο της Γέννα η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα και ζητά συγγνώμη γιατί α, βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ σήμερα. Στο 20ο αιώνα, λοιπόν, οι πιο πολλοί κανόνες του Διεθνούς Εθνικού Δικαίου, PIL, ε, ορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Μόνο στο τέλη της δεκαετίας του 90 τα κράτη-μέλη δώσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο με πολύ σημαντικά νομοθετήματα. Ωστόσο, αυτή η Ευρωπα... του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου προκαλεί προβλήματα. Το PIL δεν κωδικοποιείται σε ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Κατανείμεται σε διάφορα νομοθετήματα, διαφορετικού νομοθετικού ε, επίπεδου. Καταρχάς έχουμε τις ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αν και ε, έχουμε εντυπωσιακό αριθμό ε, ευρωπαϊκών ε, κανονισμών, 15, και είναι πολύ καλής ποιότητας, παραμένει γεγονός ότι είναι καταναμημένη η νομοθεσία σε διάφορα νομοθετήματα και αυτό μας ανησυχεί. Καταρχάς, οι τρέχοντες κανονισμοί δεν τελικά παρτίζουν ένα συνεκτικό σύνολο και εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιοι τομεί του διεθνού δικαίου, το, οι οποίοι δεν πραγματεύονται πουθενά, όπω το εταιρικό δίκαιο. Και το θέμα, για παράδειγμα, της δικαιοδοσία, το θέμα της παραβίασης δικαιωμάτων προσωπικού. Και εκεί λοιπόν εξαρτώμαστε από άλλες πηγές δικαίου. Κατά δεύτερον, το ιδιωτικό διεθνές δικαίου ως ε, σύνολο δεν ε, εξαρτάται από συγκεκριμένους κανόνες ε, που έχουν να κάνουν μόνο για παράδειγμα με τα συμβάσεις και το διαζύγιο. Όχι, περιλαμβάνει και ένα γενικό τμήμα που περιλαμβάνει νομικές διατάξεις και αποφασίζει το πόσο αποδοτικό και αποτελεσματικό είναι αυτό το δίκαιο. Και εδώ λοιπόν έχουμε κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα διπλή υπηκότητα, για παράδειγμα, όταν υπάρχει θέμα ηθαγένειας. Δεν ε, υπάρχει απάντηση στα θέματα αυτά από τους κανονισμούς και ε, αυτό τελικά καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία κατά βούληση. Ύστερα έχουμε τις διεθνείς συμβάσεις οι οποίες ε, και είναι πιο σημαντικές και υπερέχουν του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεύτερο θέμα, που μας παρουσιάζει πρόβλημα. Έχουμε κάποιες αλληλαπικαλύψεις, για παράδειγμα οι δημόσιες πολιτικές, το κράτος δικαίου, σε ό,τι αφορά ε, προβλήματα με την Ισπανία, με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε κανονισμός λοιπόν περιλαμβάνει κανόνες για τέτοιες αρχές. Προφανώς όμως τέτοια ζητήματα ε, ρυθμίζονται ξανά και ξανά και έτσι υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και έτσι Αυτές οι αλληλεκαλύψεις προκαλούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όταν δεν υπάρχει εναρμόνιση, για παράδειγμα, για την ελεύθερη επιλογή δικαίου. Ε, διαφέρουν πολύ οι κανόνες στον πρώτο και δεύτερο κανονισμό και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις αρχές ε, του Δυτικού Διεθνούς Δικαίου. Αυτές οι ανησυχίες λοιπόν έχουν οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας ομογενής ευρωπαϊκός κώδικας για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Το 2010 ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ελπίδα και παραθέτω ο απότερος σκοπός της νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μια συνεκτική κωδικοποίηση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Τέλος παράθεση. Το Μάρτιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ατζέντα για τη Δικαιοσύνη για το 2020 ανέφερε και παραθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η κωδικοποίηση του υφιστάμενου δικαίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στους τομείς σύγκρουσης τη νομοθεσία. Η κωδικοποίηση συνήθω εννοείται ω ε, μια συστηματική καταγραφή ενός συνολικού νομοθετικού κλάδου σε ένα και μόνο νομοθέτημα. Η κωδικοποίηση αυτή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανεξάρτητα, μάλλον ανάλογα με το πώς ορίζεται το νομικό ζήτημα. Έχουμε το θέμα της επιλογής του δικαίου, του ισχυντός δικαίου και τους διεθνούς δικαιοδοσίας. Αν ε, θα κοιτάξουμε για παράδειγμα αυτά τα δύο, δύο διαφορετικούς τομείς, η κωδικοποίηση θα περιοριστεί σε άλλους τομείς και ουσιαστικά θα παρατηρηθούν δύο κώδικες. Να κοιτάξουμε τώρα τα πλέον εκτήματα μιας κωδικοποίησης ενδεχομένω. Η πρώτη, το πρώτο όφελος, το πρώτο πλέον έκτημα, ορατότητα. Δυνατότητα επισκόπησης. Ένας ευρωπαϊκός κώδικας θα μπορούσε να δημιουργήσει και μια άλλη αντίληψη σε τρίτα κράτη και να οδηγήσει σε σύγκληση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου τρίτων κρατών και έτσι να οδηγήσει σε μια πιο παγκόσμια εναρμόνιση στη λήψη αποφάσεων κατά δεύτερον. Ένας ενιαίος ιδιωτικός κώδικας μπορεί να επιτρέψει καλύτερη εφαρμογή στην πράξη γιατί θα είναι πιο προσβάσιμος ο κώδικας τρίτον ευρωπαϊκή κωδικοποίηση θα αποτελούσε μια εξαιρετική ευκαιρία για να καλυφθούν τα χάσματα στο τρέχον ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Αλλά ούτε καν μια κωδικοποίηση δεν θα μπορούσε να καλύψει όλους τους νομικούς τομείς, γιατί θα ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συνένεση σε κάποια πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως ε, για παράδειγμα η παραβίαση των δικαιωμάτων του προσωπικού και το καθεξής. Επίσης, πολλά κράτη-μέλη είναι ήδη μέρη και έχουν προσυπογράψει διεθνεί συμβάσει, τις οποίε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μονομερό να αποκηρύξει. Τέλο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενό Ευρωπαϊκού Κώδικα θα ήταν ότι αν υπάρχουν ε, επικαλύψεις ή αντουκριόμενες ε, νομοθεσίες, αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με την εισαγωγή ενός γενικού τμήματος και η κωδικοποίηση επίσης των γενικών αρχών θα έπρεπε να αφήνει περιθώριο για πιο ε, λεπτομερείς διευκρινήσεις στους διάφορους νομικούς τομείς. Παρά όλα αυτά τα πλανεκτήματα, μια κωδικοποίηση αναπόφευκτα θα αντιμετώπιζε και πολλά εμπόδια. Καταρχάς, δεν υπάρχει σήμερα νομοθετική αρμοδιότητα για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό κώδικα για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ακούσαμε πριν από λίγο από τον Αντιπρόεδρο κάποια λόγια σε ό,τι αφορά το Γενικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και του Γενικών Διαδικασιών για το οικογένειακό Δίκαιο. Άρα θα έπρεπε να συμμορφωθούμε σε μια γενικότερη νομοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα είδη και επίση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιε ειδικέ πτυχέ του οικογενειακού δικαίου. Άρα η κωδικοποίηση των γενικών αρχών του ιδιωτικού διεθνού δικαίου που θα πρέπει να καλύψει και του δύο τομεί, μα παρουσιάζει πολύ σοβαρά τεχνικά και νομικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά οξύνονται με, από την Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία σε, και τις ιδιαίτερες στάσεις που έχουν σε ό,τι αφορά την δικαστική συνεργασία. Τέλος. Έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τον ε, τρίτο κανονισμό που ισχύει σε 16 κράτη-μέλη και ε, ο κανονισμός Ρώμη 3, συγγνώμη, μας παρουσιάζει προβλήματα γιατί έχουν, έχει επικυρωθεί μόνο από 16 κράτη-μέλη και πόσα ήταν η αντίδραση των άλλων κρατών μέλων που δεν έχουν προσυπογράψει. Επίσης, επί υπάρχουν και άλλα εμπόδια προς κόμματα σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει δικαστική εμπειρία για την εφαρμογή του, του κώδικα αυτό. Άρα, μια συνεκτική κωδικοποίηση θα μπορούσε να επιλύσει πολλά προβλήματα και κυρίως να υπάρχει καλύτερη επισκόπηση και συνοχή και πρόσβαση. Ωστόσο, υπάρχουν και σοβαρά θεσμικά προσκόμματα και αυτά καθιστούν μάλλον ε, απίθανο το να πραγματοποιηθεί αυτό στο εγγύ μέλλον. Ο Ευρωπαϊκό Κώδικα, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ενώπιον μας. Θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε πιο τομεακέ κωδικοποίησει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το συμβατικό δίκαιο, το συζυγικό δίκαιο. Με μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάποιες ε, να επιλύσουμε κάποια από τα προβλήματα και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία θα μπορούσαν να αποφασίσουν κατά περίπτωση κατά πόσο θα κανουν οπτήν ή όχι. Ύστερα, τομεακή κωδικοποίηση θα σήμαινε κατά πάσα πιθανότητα λιγότερη αντίσταση. Ο τρίτος τρόπος για το μέλλον. Κωδικοποίηση περιορισμένη σε κάποιους συγκεκριμένου τομεί του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Κανονισμός Ρώμη 0, όπως αναφέρεται. Ωστόσο, αυτό θα προκαλούσε τα ίδια προσκόμματα και εμπόδια όπως και μια γενικότερη κωδικοποίηση των γενικότερων αρχών. Άρα, συνοψίζοντας, όλες οι προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας έχουν πλανεκτήματα και μειονεκτήματα. Προτείνουμε μια σταδιακή προσέγγιση μια σταδιακή κωδικοποίηση του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου με τρεις πυλώνες, ένα μοντέλο με τρεις πυλώνες, το οποίο σταδιακά θα μας δώσει ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο και το οποίο μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να οδηγήσει σε έναν ευρωπαϊκό κώδικα. Στον πρώτο πυλώνα του μοντέλου αυτού συστήνουμε μέτρα για να συμπληρωθεί το τρέχον και εκτιμένο να πληρωθούν τα χάσματα του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου που ανέφερα Επίσης να υποστηρίξουμε προσπάθειες για αρμονισμένους κανόνες για την εφαρμογή του δικαίου αυτού. Στο δεύτερο πυλώνα τώρα συστήνουμε νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν το κεκτωμένο στο διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Δηλαδή να συνενώσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία να είναι πιο ομογενής η εφαρμογή αλλά και η σχεδιασμός. Ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος περιγράφεται λεπτόμερος περιλαμβάνει μέτρα για να βελτιωθεί το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως η ίδρυση ομάδας κεκτημένου για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Η πρόεδρος. Θα μπορούσατε, αν θέλετε, να ολοκληρώσετε. Ναι, ναι, ναι, ναι τελευταία σελίδα, τελευταία σελίδα. Για να παρακολουθήσουμε λοιπόν την εφαρμογή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην πράξη δημιουργώντας ειδικά δικαστήρια για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων ευρωπαϊκή για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, προκειμένου να υπάρχει και πρόσβαση για τους επαγγελματίες στην ε, νομολογία και τέλος βελτίωση της γενικότερη νομική εκπαίδευση και κατάρτιση των δικαστών στον τομέα του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Διεθνής Δικαίου. Σε... Συνοψίζοντας, προτείνουμε να αναβληθούν τα μέτρα για ε, έναν συνεκτικό κώδικα στην παρούσα φάση και προτείνουμε ένα μοντέλο τριών πυλώνων που σταδιακά θα βελτιώσει θεσμική ομοιογένεια για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και ενδεχομένως μακροπρόθεσμα να προλυάνει το έδαφος για έναν συνεκτικό ευρωπαϊκό κώδικα. Ευχαριστώ καθηγητά Φανχάιν. Ήσασταν λίγο ξεπεράσατε το χρονικό όριο, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και πάρα αυτά θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Να καλωσορίσω λοιπόν ε, εδώ τον καθηγητή Πιερ Καλέ από το Παρίσι το Πανεπιστήμιο Παρίσι Σουτ και τον κύριο Μάικλ Κλάνσι, δικηγόρο από την ε, Law Society of Scotland. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο σκοπεύει να πάρει το λόγο πρώτος. Ο καθηγητής Καλέ Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με προσκαλέσατε στο σημερινό εργαστήρι. Θα ήθελα να συζητήσουμε την απλούστευση του κανονισμού για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Είναι τρεις οι άξονες ε, θα επικεντρωθώ στους δύο βασικούς. Ε, η κατάργηση ε, της ανάγκης επιστοποίησης και το πολύγλωσσο έντυπο. Για την επικύρωση των εγγράφων, ε, ο στόχος είναι να εγκαταστούν αυθεντικά τα έγγραφα όταν, παραδείγματος χάρη, έχουμε ε, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο και θέλουμε να αναγνωριστεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, χρειάζεται η επικύρωση ε, που συνεπάγεται μια μακρά διαδικασία. Αυτό Όμω δεν υπάρχει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι έχουν προσχωρήσει τα κράτη-μέλη στη Σύμβαση της Χαγή και η επικύρωση αντικαθίσταται από μια απλουστευμένη διαδικασία ε, της φραγίδα της Χαγή. Αυτό μπορεί να έχει ένα κειμενόμενο κόστος ε, ανάλογα με το κράτος ε, από 0 έως 50 ευρώ κοστίζει η σφραγίδα της Χάγης ανάλογα με το κράτος μέλος. Η πρόταση κανονισμού λοιπόν έγινε στην κατάργηση της επικύρωσης και της φραγίδας της Χάγης για την, ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι η κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης ήδη έχει ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όταν μιλάμε για αυθεντικά δημόσια, γνήσια δημόσια έγγραφα. Ε, όλες, όλοι οι κανονισμοί των Βρυξελών 1 και 2 προβλέπουν στο πεδίο εφαρμογής τους ότι δεν χρειάζεται ε, καμία επικύρωση. κατάργηση λοιπόν αυτής της υποχρέωσης προκύπτει και από διεθνείς συμβάσεις ε, που έχουν υπογράψει τα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη ε, το 87 υπεγράφει μια σύμβαση των Βρυξελών ή υπήρξε και μια σύμβαση για το αστικό δίκαιο 16 2-16-17 με διάφορες συμβάσεις που μέσω κάποιων νομικών πράξεων προβλέπουν την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης. Βλέπουμε ότι μερικώς ε, ε, έχει καταργηθεί η επικύρωση και επίσης συνειδητοποιούμε ότι ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ομοιόμορφα προσχωρήσει σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που διέπουν αυτό το ζήτημα. Οπότε τι γίνεται στην πράξη όταν πρέπει να εκδοθεί ένα δημόσιο έγγραφο σε ένα άλλο κράτος μέλος, πρέπει ο πολίτης να πάει να δει αν είναι εφαρμοστέο ε, ένα νομοθέτημα που επίσης πρέπει να είναι εφαρμοστέο στο κράτος το οποίο θα χρησιμοποιήσει τον δημόσιο έγγραφο που θέλει να... Ε, παράδειγμα, ε, είμαστε στη Γαλλία και διαπιστώνουμε ο πολίτης εάν στην Ιταλία, ή στην Ελλάδα ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί χρειάζεται να ε, φέρει την σφραγίδα της Χάγης, παραδείγματο χάρη στη Γαλλία. Και ο λόγος είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν προσχωρήσει στις ίδιες συμβάσεις. Οπότε ο κανονισμός γενικεύει την κατάργηση της επικύρωσης και αυτό με ισχύει στην επικράτεια όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικότατη η πρόοδο διότι έτσι διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή ζωή των πολιτών που χρειάζονται, παραδείγματο χάρη, ε, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ε, στη χώρα όπου διαμένουν, αποφεύγοντας και το κόστος που σε ορισμένες φορές ε, είναι οριακό ή πολύ χαμηλό για τη σφραγίδα της Χάγης. Έτσι καταργείται αυτό το κόστος και κυρίως κερδίζουμε χρόνο, κερδίζει χρόνο ο πολίτης ε, για την έκδοση του δημοσίου εγγράφου. Ποιος κίνδυνος ελοχεύει με την κατάργηση της ανάγκης επικύρωσης πολλαπλασιασμού των πλαστών εγγράφων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ο στόχος ήταν να επιστοποιηθεί η γνησιότητα του έγγραφου. Αυτός ο κίνδυνος όμως δεν φαίνεται υπαρκτός ε, για δύο λόγους. Όπως σας είπα, η κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη έχει ήδη ξεκινήσει για διάφορα έγγραφα και ανάμεσα στις, σχέσεις, στις διμερείς σχέσεις ορισμένων ε, κρατών μελών. Και όπου έχει αυτό συμβεί δεν παρουσιάστηκε αύξηση των πλαστών εγγράφων ε, που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η σύμβαση της σφραγίδας της Χάγης ε, πολύ αμφιβάλλουμε αν καταπολεμά την ε, απάτη τελικά <coughs> διότι σε τι βασιζόταν ε, η καταπολέμηση απάτης το ότι βάσει των διατάξεων για την σφραγίδα της Χάγης υπάρχει ένα μητρό, ένα κοινό μητρό και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξακριβώσουμε σε αυτό το Μητρό αν έχει όντως εκδοθεί αυτό το έγγραφο. Όμως, λίγοι, πάρα πολύ λίγοι ε, πηγαίνουν και συμβουλεύονται αυτό το Μητρό των εγγράφων που φέρουν την σφραγίδα της Χάγης. Ε, για τον εντοπισμό τώρα των πλαστών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνουμε έναν ελεγκτικό μηχανισμό που ε, δράζεται επί της διοικητικής συνεργασίας ε, αν συντρέχει εύλογη υποψία ε, και προβλέπεται και η δημιουργία μιας κεντρικής αρχής στην οποία θα προτείνονται όλοι για να εξακριβώσουν τη γνησιότητα ενό εγγράφου εάν λειτουργήσει αισίως αυτή η διοικητική συνεργασία με πολύ αποτελεσματικό τρόπο θα καταπολεμήσουμε την απαραίτηση τη μεταγνήση έγγραφα, διότι ξαναλέω οι αρχές που έχουν λάβει ένα έγγραφο που φέρει την ε, Ασφαλεία της Χάγης πολύ σπάνια συμβουλεύονται το σχετικό μητρό. Υπάρχουν ε, όμως ε, δύο ε, ανησυχίες. Πρώτον, σε σχέση με το ουσιαστικό δίκαιο για τον δημόσιο κατάλογο των εγγράφων, πάντοτε θα έχουμε κάποια έγγραφα που δεν καταχωρίζονται σε αυτόν τον κατάλογο. Οπότε είναι απλούστερο να μην έχουμε ένα κατάλογο και να καλύπτουμε όλες τις αποφάσεις εγγνής, έγγραφα, αποφάσεις, διαταγές, έγγραφα αστικού δικαίου, διότι αν δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά τα έγγραφα μέσα στον κανονισμό, ε, δεν θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση της επικύρωσης παρά μόνο εάν προβλέπονται σε κάποιο άλλο κανονισμό. Για ένα έγγραφο που σχετίζεται με τη Διαθήκη, παραδείγματο χάρη, ε, θα προβλέπεται αυτό στον κανονισμό που ε, διέπει τις διαθήκες σε αντίθετη περίπτωση δεν θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση επικύρωσης ε, ε, Τέλο πάντων, θα ήταν απλούστερο να μην έχουμε κανένα κατάλογο, θα ήταν απλούστερο να το έχουμε προβλέψει για όλα τα δημόσια έγγραφα. Και δεύτερη ανησυχία υπάρχει ο κανονισμό των Βρυξελών για τι αποφάσει και τα γνήσια έγγραφα. Σε, μέσα σε αυτόν τον κανονισμό δεν υπάρχει καμία ναι. διαδικασία χάρη στην οποία θα μπορούσε μια αρχή που αμφιβάλλει για την γνησιότητα μια δικαστική απόφαση ενό δημοσίου εγγράφου για να προβεί σε έναν έλεγχο σε μία εξακρίβωση θα μπορούσαμε ε, να φανταστούμε ε, ε, αυτήν την διάταξη να διευρύνεται σε όλους τους κανονισμούς που αφορούν σε όλα τα υπόλοιπα δημόσια έγγραφα, αλλά αυτό δεν έγινε δυστυχώς. Ε, εν συντομία θα ήθελα να σχολιάσω τώρα το δεύτερο άξονα, δηλαδή τα πολύγλωσσα έντυπα για τη γέννηση, για το θάνατο, για, την, για τις καταχωρισμένες εταιρικές σχέσεις, για τους γάμους και το καθεξής. Ε, είναι ε, μια εναλλακτική λύση για τα δημόσια έγγραφα που κυκλοφορούν στα κράτη-μέλη και βάσει αιτήματο ε, του πολίτη θα εκδίδονται. Δηλαδή θα είναι ένα ισοδύναμο, αν θέλετε, έγγραφος προς το δημόσιο, επίσημο δημόσιο έγγραφο. Ε, με, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου ε, ουσιαστικά εξυπηρετούμε τον ίδιο στόχο. Δεν αντικαθίσταται το επίσημο δημόσιο έγγραφο για την ε, κληρονομική διαδοχή, αλλά είναι ένα επιπρόσθετο ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, ένα επιπρόσθετο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Ο στόχος των πολύγλωσσων εντύπων είναι να ε, απαλληφθεί το πρόβλημα της μετάφρασης των εγγράφων με την ενοποίηση δε οι αναφορές ε, που γίνονται στο έγγραφο είναι σαφέστερες και αποφεύγουμε έτσι προβλήματα κατανόησης διότι ε, κάθε ένωμη τάξη προβλέπει άλλες αναφορές στα δημόσια έγγραφα και μπορεί ναι, κάποιο κράτος να μην κατανοεί τις αναφορές που βρίσκει σε ένα δημόσιο έγγραφο άλλου κράτους. Ε, ποια ζητήματα τίθενται και αυτά προβλέπονται και στην πρόταση. Ότι πρέπει να παραμείνουν προαιρετικά αυτά τα πολύγλωσσα έντυπα. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Θα πρέπει να διαφυλαχθεί η δυνατότητα κυκλοφορία των επισήμων δημοσίων εγγράφων, διότι απηχούν και τι ιδιαιτερότητε των ε, οικείων νομικών συστημάτων και αυτή είναι η κυλομορφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κλείσω τώρα ε, λέγοντα ότι το νόημα αυτών των ε, πολύγλωσσων εντύπων είναι ε, η σχέση τους με την πράξη, η ληξιαρχική πράξη ε, γέννησης, θανάτου, απόσπασμα ποινικού μητρώου. <clears throat> δηλαδή, η διατύπωση έχει ε, καταλητική σημασία για να ε, καταλάβουμε αν συνενεί ε, αυτός του οποίου εκδίδεται το έγγραφο και έχω την εντύπωση ότι μια τέτοια ανησυχία υπήρχε στην Γαλλία. Δεν είναι τίποτα το αρνητικό αυτή η εξέλιξη για τα πολύγλωσσα έντυπα, όμως στο βαθμό που δεν θα ε, γενικευθεί η χρήση τους ε, και ε, που ο στόχος τους θα είναι μόνο να αποδείξουν ένα γεγονός όπως η γέννηση, θάνατος κτλ. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε καθηγητά Καλέ. Σχεδόν τηρήσατε και το χρόνο που σας αναλογούσε. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κλάνση, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μου χαρά ε, ήρθα εδώ στο φόρουμ για το αστικό δίκαιο και τη δικαιοσύνη για να δούμε πώς θα είναι πιο εύκολη η ζωή των Ευρωπαίων. Γιατί αυτό είναι ο στόχος των συνθήκων. Για να δούμε το ότι δεν πρόκειται μόνο για υποχρέωση που προκύπτει μέσω της συνθήκης αλλά είναι και κάτι τελείως λογικό. Όντως υπήρχε κάθε καλή πρόθεση με τον κανονισμό του 2013-2028. Εκεί όπου είχαμε αυτή την νομοθετική πρόταση για να σταματήσει η γραφειοκρατία όσον αφορά την επικύρωση. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα για να ε, υπάρχει πιο απλή νομοθεσία, όπως είπε ο καθηγητής Καλέ. Ήδη έχει προχωρήσει σε πολλούς τομείς του δικαίου αυτή η πρωτοβουλία. Για να δούμε πώς θα έχουμε ελεύθερη ε, διαβίβαση των εγγράφων. Και τελικά το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προέβη αυτή την ε, πρόταση κανονισμού που σήμερα εξετάζουμε. Για να λάβουμε υπόψη τι έγινε στην σύμβαση του 69 της Χάγης. Εκεί που καταργήθηκε το προαπαιτούμενο της επικύρωσης των δημοσίων εγγράφων. Επρόκειτο για τον τύπο ε, μέσω του οποίου τα προξενία ε, ή οι πρεσβείες ε, επικύρωναν το έγγραφο αναγνωρίζοντας την υπογραφή, την ιδιότητα του προσώπου που επέγραφε κλπ. Οπότε με αυτή τη σύμβαση, αντί για όλη εκείνη την διαδικασία επικύρωσης, έχουμε τώρα τη σφραγίδα της Χάγης. Ε, οπότε έχουμε τώρα τα έγγραφα τα οποία αναγνωρίζονται από ένα άλλο κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εξεδόθησαν. Και είπαμε τώρα ότι έχουμε επίσης κάποια επίσημα δημοσιέγγραφα που έχουν σχέση με δικαστήρια. Δηλαδή πρόκειται για αποφάσεις για συμβολογραφικές πράξεις και άλλου είδους πιστοποιητικά ε, ε, για πιστοποιητικά θανάτου, αποσπάσματα εμπορικών μητρών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. Και είχαμε επομένως 12 κατηγορίες όπως ε, οικογενικής κατάστασης, πιστοποιητικά, απόσπασμα ποινικού μητρώου, αλλά δεν Τότε, σύμφωνα με την πρόταση αυτή τα ιδιωτικά έγγραφα. Πάντως είπαμε ότι θα υπάρχει τώρα μια ρήτρα διαφύλαξης του πίν κατά των πλαστών εγγράφων. Είπαμε ότι όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την γνησιότητα του εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κρατημέλη μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από το κράτο μέλο έκδοση του εγγράφου. μπορούν απευθείας να απευθυνθούν επομένως στο άλλο κράτος μέλος. Στο άρθρο 11 έχουμε ε, τα έντυπα, τα καθιερωμένα, τα πολύγλωσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε εδώ πέρα διάφορες, ε, ε, διάφορες τυπικότητες και είπαμε ότι τώρα προσπαθούν οι ε, οι αρχές να φέρουν λιγότερη γραφειοκρατία. Πρόκειται για κάποιους ε, στόχους ε, ούτω ώστε να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τη ελεύθερη διακίνηση οι πολίτε, να έχουν λιγότερο κόστο, λιγότερη γραφειοκρατία. Και σύμφωνα με. Την πρόταση αυτή έγιναν κάποιε προτάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, διευρυνθεί το πεδίο των δημόσιων εγγράφων, να περιλαμβηθεί για παράδειγμα και το θέμα της μετανάστευσης, το θέμα του ποινικού μητρώου σε άλλους τομείς ε, της ε, ατζέντα για την ε, δικαιοσύνη και την ασφάλεια και επίσης να προσθεθεί και ένα πολύ γλωσσό φόρουμ για τα ονόματα, για το αν κανείς είναι πατρεμένος ή όχι κτλ. Και η σχετική ομάδα έχει εξετάσει την πρόταση από τον Απρίλιο του 2013 και μία πλειοψηφία των κρατών μελών δεν αποδέχτηκε το πεδίο εφαρμογή του αρχικού κειμένου όπω το παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όπω το τροποποίησε το Κοινοβούλιο. Και η Ιταλική Προεδρία λοιπόν πρότεινε να, να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογή στο. στην οικογενειακή κατάσταση για να ισχύει μόνο για την γέννηση, θάνατο, όνομα, γάμους, ε, καταχωρισμένη ε, σχέση, ε, υιοθεσία, παιδιά, κατοικία, ηθαγένεια και υπηκότητα. Η Ιταλική Προεδρία πρότεινε και μία λύση για τα πολύ φόρουμ, για τις τα γλωσσα έντυπα. Και η απλοποίηση της αποδοχής των εγγράφων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμβάλλει στην συμπλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδιαίτερα σε θέματα ταυτότητας. Γιατί πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα βασικό, όπως είναι και το θέμα γέννησης θανάτου, κατοικίας, γάμου, διαζυγίου, εκπαίδευσης και ενδεχόμενος να ωφεληθούν και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αν συμπεριληφθούν στο μέλλον καταχωρισμένα εταιρικά έγγραφα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόταση που εξετάζουμε στην παρούσα φάση. Το μειονέκτημα είναι ότι υπάρχουν ανησυχίες για το κόστος ενδεχομένω για την επαλήθευση αμφίβολων εγγράφων και φυσικά όσο πιο ευρύ το πεδίο εφαρμογή, τόσο πιο πολλές ενδεχομένως να είναι οι ενστάσεις και οι εξετάσεις αυτές. Αλλά σίγουρα υπάρχει πλέον να υπάρχει ένα μετριοπαθές πρόγραμμα όπως αυτό που προτείνει η Ιταλική Προεδρία με μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογή όταν έχει εγκαθιδρυθεί σωστά το σύστημα και ακούσαμε την ιδέα αυτή σήμερα το πρωί. Το άρθρο 21 προβλέπει μια αναθεώρηση κάθε τρία χρόνια που περιλαμβάνει ε, το κατά πόσο θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τι θα σημαίνει αυτό ακριβώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο στην παρούσα φάση εκδίδεται 400.000 αποστήλες ε, σφραγίδες της Χάγης ανά έτος, αλλά μόνο το 25.000 θα ήταν ενδεχομένω στο πεδίο εφαρμογή τη πρόταση. Ε, για άλλε χώρε αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλο ω αριθμό και ήταν δύσκολο να κάνουμε την εκτίμηση για τις πολύγλωσσες ε, φόρμες, τα πολύγλωσσα έντυπα. Δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για να ξέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο τέτοια έντυπα για χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα πλέον πλεονεκτήματα για να δούμε τι σημαίνει ένα τέτοιο έντυπο στη διαδικασία και στα διαδικαστικά και στην εκπαιρέωση κάθε κράτους μέλους. Δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη να υπάρξει ε, ευρωπαϊκή έκδοση των εθνικών εγγράφων οικογενειακής κατάστασης. Ένα μειονέκτημα το οποίο έχω διαπιστώσει αλλά μου αρέσει είναι ότι έχουν και παιδεία μεταφρασμένα και μη μεταφρασμένα τα οποία απλά μεταγράφονται από το αρχικό εθνικό έγγραφο. Ίσως το μεταγεγραμμένο κομμάτι θα έπρεπε να καταργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τα βασικά γεγονότα στην ε, πολύγλωση έκδοση. Θα ήταν και πιο γρήγορο και πιο φτηνό κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι μόνο πλεονεκτήματα έχει. Χρειάζεται μια πιο σαφή σχέση μεταξύ της πρότασης αυτής και της ατζέντα για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Η πρόταση για μια ηλεκτρονική ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πιο στενά τον κανονισμό για να δούμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκληθούν προβλήματα εφαρμογής του κανονισμού σε ό,τι αφορά την ε, ηλεκτρονική αγορά. Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής ε, θα επιτρέψει την τεχνική εξέταση καταρχάς των προτάσεων και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν επαρκέ ε, χρονικό διάστημα για να το πράξουν αυτό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κανονισμό ενδεχομένω να βοηθήσει να ενοποιηθεί η αγορά καταργώντας τα, προσκόμματα, αλλά παράλληλα θα δώσει προτίμηση στις, ε, στους και όχι στις επιχειρήσεις και θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες πτυχές πριν ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και όπως λέει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2004 για την αγωνιστικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως να αποτελέσει εμπόδιο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Ίσως λοιπόν το Κοινοβούλιο καλά θα έκανε να εξετάσει περαιτέρω εργασίες στον κλάδο αυτό παράλληλες για να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε όλα τα εμπόδια τα οποία υφίστανται στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριε. Ευχαριστώ κύριε Κλάνση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση του φακέλου αυτού. Όπως ξέρετε, είμαι συγγητρία για τα δημόσια έγγραφα και κληρονόμησα αυτό το φάκελο, αυτό το θέμα από το κύριο Ραπκάη και θεώρησα στην αρχή ότι ήταν αρκετά προφανές ότι θέλουμε να προωθήσουμε την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών και των επιχειρήσεων αποτελεί ένα κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίστευα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση της επικύρωσης, ε, της φραγίδας της Χάγης, ε, εισαγωγή της ε, πολύγλωσσης ε, μορφής, η απλοποίηση της μετάφρασης και η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών μελών. Θεωρούσα, εν πάση περιπτώσει, ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε πολύ γρήγορα να συμφωνηθεί μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Εξαιρετική δουλειά έχει κάνει ο κ. Ραπκάη, γιατί το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2013 έχει εγκρίνει μια κοινή τοποθέτηση πάνω από ένα χρόνο δηλαδή, και το Κοινοβούλιο ενίσχυσε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύξησε τον αριθμό των δημοσίων εγγράφων που θα υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, εισήγαγε Επιπρόσθετες, επιπρόσθετα πολύγλωσσα έντυπα περιόρισε την ανάγκη για επικοινωνμένες μεταφράσεις και μεταφέρθηκε το κόστος μετάφρασης από τον πολίτη στην ε, δίκηση, στις υπηρεσίες. Αυτή η τελευταία πρόταση του να μεταφερθεί το κόστος στις δημόσιες υπηρεσίες, φαντάζομαι ότι αυτή η πρόταση λοιπόν δεν θα ήταν και τόσο δημοφιλής στα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ, ανακάλυψα ότι το Συμβούλιο είναι πολύ πολύ διστακτικό. Η Ιταλική Προεδρία το είχε βάλει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, προσπάθησε να πετύχει συμφωνία, δεν τα κατάφερε. Ελπίζω η Ελληνική Προεδρία να καταφέρει να ολοκληρώσει το θέμα αυτό, όπως και μας είπε και η κυρία Λίμπινα Εκπέ. Είναι ελπίδα και της Λιτωνικής Προεδρίας. Επάς θα είναι περιορισμένο στο τομέα εφαρμογή του κανονισμού. Η συζήτηση για τη μετάφραση εξακολουθεί να διεξάγεται. Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί Ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει τριμερής διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Εγώ και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ανοίξουμε τη συζήτηση, να θέσουμε ερωτήσει προς τους ομιλητές μου. Εγώ λοιπόν ρωτιέμαι το εξή και αυτό διαρωτώ με. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. δεν εμπιστεύονται τη δημόσια διοίκηση άλλων κρατών μελών. Αναφερθήκατε ότι, στο ότι πολλά κρατημέλη αναγνωρίζουν την αναγκή απλούστευσης. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και σε συμβάσεις, συνθήκες για την κατάργηση, για παράδειγμα, της επικύρωσης, της ε, αποστήλης, της φραγίδας της Χάγης και υπάρχουν ε, γλωσσά έντυπα τα οποία τα πραγματεύεται και συνθήκη για το οικογενειακό καθεστώς. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί είναι τόσο δύσκολο να σημειωθεί πρόοδος, γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε τη ζωή των πολιτών. Που ζουν ή συναλλάσσονται διασυνοριακά. Και εν πάση περιπτώσει αν ναι, το παιδιά εφαρμογή περιορίζεται στην οικογενειακή κατάσταση, όλο το θέμα των επιχειρήσεων δεν συμπεριλαμβάνεται. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ίσως έχετε και ερωτήσεις προς τους ομιλητές μας. Σας καλώ Ο κύριος Τσούκερ ζητάει το λόγο από τη Ρουμανία. Δεν ξέρω αν σωστά προσφέρω. Ο κύριος Λεμπρετό, αλλά από το κύριο Τσούκερ. Είστε Ναι, ναι, σωστά το προφέρατε, λέει. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε δώσατε το λόγο, ευχαριστούμε για τις εισηγήσεις, για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Πάρα πολύ χρήσιμα είναι. Βεβαίω όλοι μας και εγώ ίδιο θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία έχει κάνει μια διαδρομή και θα πρέπει κάποια στιγμή να επιδέχεται κάποια, κάποιον εξυγχρονισμό, κάποια επικαιροποίηση, να είναι πιο χρήσιμη. Τέλος πάντων να μην ξεχνούμε ότι έχουμε εδώ πέρα πολλές απόψεις του ζητήματος. Είπαμε ότι δεν γίνεται πλέον διασταύρωση στοιχείων όταν έχουμε ζητήματα σφαγίδας της Χάγης. Υπάρχει επομένω ε, εμπιστοσύνη. Άρα το σύστημα λειτουργεί. Να το εξυγχρονίσουμε, αλλά λειτουργεί. Αποδίδει. Δηλαδή, αν πούμε ότι οι επαληθεύσει και η διασταύρωση στοιχείων γίνεται για κάποιε περιπτώσει ότι ε, όταν ένα υπάλληλο ε, θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι αμφιβολιών, ε, τότε ο αρμόδιος αυτός υπάλληλο, όταν έρθει η ώρα να εξετάσει ένα έγγραφο και έχει αμφιβολία και λέει ότι μπορεί να είναι πλαστό, τότε, τότε αποδίδονται ευθύνες. Όπως επίσης υφίσταται τις συνέπειες και ο ίδιο ο ο οποίο χρησιμοποίησε έγγραφο το οποίο δεν είχε περάσει από διασταύρωση και επαλήθευση. Επομένως, όταν γίνεται η εξέταση του εγγράφου, τότε θα πρέπει η χειριστές υπάλληλοι να προβαίνουν σε αυτήν την επαλήθευση του αν το έγγραφο είναι πλαστό ή όχι. Αλλιώς φέρουν και εκείνη ευθύνη. Γιατί ακριβώς υπάρχει τρόπος διαπίστωσης γνησιότητος και δεν την χρησιμοποίησαν. Πώς θα γίνει τώρα όμως. Εάν έχει αμφιβολίες κάποιος υπάλληλο, θα απευθύνεται στην ε, ξένη εκδούσα αρχή και τι θα κάνει εκείνη η αρχή του άλλου κράτους μέλους. Δηλαδή ο υπάλληλο ή η υπηρεσία του θα απευθύνεται στην αρχή που εξέδωσε τον έγγραφο. Δεν έχω καταλάβει καλά. Είπαμε ότι θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Γιατί τελικά περί της γνησιόντος του εγγράφου θα αποφανθεί η αρχή που το εξέδωσε, υποτίθεται ότι το εξέδωσε. Τι θέλω να σας πω. Όχι. Δεν είναι άστοχη η προσπάθεια ρύθμισης τώρα. Απλώς θέλουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Θέλουμε αυτοί που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τη ρύθμιση αυτή να έχουν εύκολη πρόσβαση. Να μην πληρώνει τις φαγητές χάγης ο πολίτης ούτε για το κόστος της ε, επικύρωσης. και αναλαμβάνει επομένω η αρχή στην οποία προσφεύγει ο πολίτη να, ε, να έρθει σε επαφή με την ε, ομόλογη αρχή στο άλλο κράτος μέλος. Να σκεφτούμε όλες τις λεπτομέρειες, τι θα γίνει με τα δικαστήρια, Φερρυπίν. Θα πρέπει να έχουμε τέτοιου προοπτική, σφαιρική, μακρόπνοια. Έτσι θα φτιάξουμε μια ρύθμιση λειτουργική. Ένας υπάλληλος ληξιαρχείου δεν έχει τα στοιχεία που χρειάζονται για να καταλήξει το αν μπροστά του βρίσκεται ένα πλαστό έγγραφο. Εκτός αν πρόκειται για περίπτωση κατάφορης ε, ε, ε αλλίωσης του εγγράφου. Σε περισσότερες περιπτώσεις πάντως δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η γνησιότητα. γιατί όταν κάποιος ε, ζημιωθεί από κάποιο πλαστό έγγραφο, τότε να ζητώνται ευθύνες και φέρει την ευθύνη και ο υπάλληλο ο οποίος θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει τη γνησιότητα. Θα πρέπει επομένω να δούμε στην πράξη τι προβλήματα προκύπτουν να επικαιροποιήσουμε τη ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις μεταβλητές. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο προλαλήσαντες. Είναι εξαιρετική η παρουσίαση που έκαναν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ε, καθηγητά Καλέ ε, διότι είχε έρθει επισκέπτης ε, στο δικό μου πανεπιστήμιο. Ήταν, όλες είχε ξεκινήσει την καριέρα του τότε, χαίρομαι που τον ξαναβλέπω. Λοιπόν, για τα πολύγλωσσα έντυπα δεν είναι απλώς πολύγλωσσα, είναι και ομοιόμορφα, ε, διότι ο τύπος τελικά επηρεάζει και την ουσία. Ε, φυσικά μπορούμε ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα αντικαταστήσουμε τα δημόσια έγγραφα σε ένα ε, πρώτο στάδιο, αλλά τελικά κάτι που λειτουργεί επιπρόσθετα στο τέλος γίνεται ο κανόνας. Αν κρίνουμε από την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα προετοιμάζονται διάφορα έγγραφα για τα πιστοποιητικά γεννήσεως, παραδείγματος χάρη. Ε, υπάρχουν θέματα ακόμη και με τη λέξη που χρησιμοποιείται σε διάφορες γλώσσες ε, για το φύλλο. Τέλος πάντων, ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, οι προσπάθειες αυτές ε, θα ε, ενισχύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, διότι ο καλύτερος τρόπος για να διευκολύνει κανείς την ελεύθερη κυκλοφορία θα ήταν να καταργήσει τα κράτη-μέλη και θα υπήρχε ένα μεγάλο κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα ήταν πάρα πολύ εύκολη η κυκλοφορία των προσώπων. Βεβαίως, αυτό που με ανησυχεί κυρία Ντελβού είναι αυτά που είπατε για τις διασυνοριακές επιχειρήσει, Δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό, με αυτή την πραγματικότητα. Ούτε επιθυμώ να αλλάξει. Όμω θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή από πλευράς εκείνων και όχι το ανάποδο, να μην προσαρμοστούν τα κράτη, αλλά οι επιχειρήσει. Καταλάβατε τι εννοώ. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή η κατεύθυνση που ακολουθούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπερτερεί ο σεβασμός ε, των εθνικών δικαίων σε σχέση ε, με τις προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σεβασμός των, ε, της ένομης τάξης με αυτή την σφραγίδα της ε, Χάγης ε, και είμαι υπέρ της διατήρησής της. Απλώς θα πρέπει να υπάρξει μια ταχύτερη διοικητική διαδικασία εξακρίβωση των στοιχείων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει. Φυσικά, αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ναι, θα πρέπει να δεχτούμε και τα μειονεκτήματα που αυτό έχει. Σας ευχαριστούμε. Ε, κύριε Μπονέ, ήσασταν ξεκάθαρος ως προς την ε, άποψη που υπερασπίζεστε ο κύριος Πούτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ όσους έκαναν αυτή την παρουσίαση. Είδαμε την εξέλιξη στο Συμβούλιο. Ο απότερος στόχος, όπως και εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι να απλοποιήσουμε την ζωή των πολιτών. Όμως, ταυτόχρονα θέλουμε να ακούσουμε από το να προτείνουμε ε, μηχανισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάσουν αρνητικά τόσοι ισχύουν. Αυτή τη στιγμή ξέρω πόσο το Συμβούλιο δεν επιθυμεί ο κανονισμός αυτός να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής του και άλλα είδη εγγράφων. Όλοι γνωρίζουμε ποια προβλήματα μπορεί να ανακύψουν σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά τα φίλτρα εξακρίβωσης ε, από πλευράς των κρατών μελών. Κοιτάξτε, η επικύρωση και η σφραγίδα της Χάγης ε, στόχο έχουν να προσφέρουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και στους πολίτες αλλά και στις αρχές ε, που χρησιμοποιούν τα εκδιδόμενα δημόσια έγγραφα. Εξακριβώνεται λοιπόν η γνησιότητά τους από ε, ένα, μια ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκλείψει αυτή η ασφάλεια σε σχέση με τα δημοτολόγια, παραδείγματος χάρη, την οικογενειακή κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία σε σχέση με τη γνησιότητα ενός δημοσίου εγγράφου. Δηλαδή, εννοώ ότι ενδεχομένως θα ανακύψουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις με ένα έγγραφο ε, που υπερβαίνουν κατά πολύ το διοικητικό άχθος της εξακρίβωσης ε, αυτού του εγγράφου. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος, θέλουμε να απλωστεύσουμε τη διαδικασία. Ναι, μεν, όμως δεν μπορούμε να εξαλείψουμε όλα αυτά τα φίλτρα ασφαλείας. Φυσικά ε, οι πολίτες δεν θέλουν να καταβάλουν ε, το κόστος της φραγίδας της ε, Χάγης. Αν τους ρωτήσετε θα σας πούνε όχι, δεν θέλουμε να αναλάβουμε αυτό το κόστος, αλλά Ταυτόχρονα πρόκειται για βασικές λειτουργίες ε, του κράτους ε, και δεν μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη διαδικασία και να μην συνειδητοποιούμε, όπως είπε και ε, ο Γάλλος συνάδελφος, τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί. βλέπω θέλει άλλος το λόγο. ή ίσως ένας από του δύο εισηγητές ε, θέλουν το λόγο να απαντήσουν στα όσα έχουν ο καθηγητά Καλέ νομίζω ότι θέλετε κάτι να προσθέσετε ναι ναι δύο λόγια ω απάντηση συμφωνώ 100% με τους ε, στόχους ότι δηλαδή η κατάργηση της επικύρωσης δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της ε, ασφάλειας και έχουμε αύξηση άλλωστε των φαινομένων πλαστών εγγράφων. Πρώτα πρώτα, έχουμε πολλά κείμενα νομοθετικά της Ένωσης που έχουν καταργήσει την διαδικασία της επικύρωσης. Όμως, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει έλεγχος. Όμως, αυτό το σχέδιο κανονισμού λέει ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει έλεγχος σε την περίπτωση που γενικεύεται η κατάργηση της επικύρωσης. Επίσης, κάποιος είπε για τη Σύμβαση της Χάγης ότι λειτουργεί καλά, ναι, αλλά ξέρετε πώς το βλέπει κανείς. Ε, χρειάζεται συστηματικό έργο, τόσο ώστε κανεί να δει το ότι θα... Ε, μπορεί, οποιο, μπορεί κανένας να, κάνει τις φραγίδες της Χάγης και στο σπίτι του με τον ε, υπολογιστή του. Α, το θέμα είναι πώς θα καταπολεμηθεί η απάτη. Παντού όλο τον κόσμο ε, κυκλοφορούν οι σφραγίδες της Χάγης και κανείς ποτέ δεν ελέγχει. Άρα πρόκειται για γενικευμένη χρήση και θα πρέπει να είναι όμως και γενικευμένη η προσπάθεια καταπολέμησης των πλαστών. Επίσης όταν έχουμε μια δημοσία αρχή η οποία έχει εύλογες αμφιβολίες για ένα έγγραφο θα επικοινωνήσει με κάποια κεντρική άλλη αρχή, η οποία θα επικοινωνήσει με την ομόλογη αρχή της ε, χώρας που εξέδωσε το έγγραφο. Όλα αυτά βεβαίω κοστίζουν. Δύσκολο να αξιολογήσουμε πόσο, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Ε, Ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρος Βαλκαρθέλ Σίζο μας είπε ότι θέλει να βρεθούν γέφυρες μεταξύ των ενόμων τάξεων και να μην έχουμε μόνο την, ε, από τα πάνω ε, η εναρμόνιση ας πούμε για τα θέματα της κοινωνικής κατάστασης. Όμως δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την εθνική νομοθεσία και η καλύτερη προστασία είναι η επικουρικότητα. Ακριβώς διότι θα πρέπει να πάνε υπόψη η εθνική νομική παράδοση. Και αυτό για όλη την Ευρώπη. Τώρα, απάτη και ευθύνη του υπαλλήλου του ελέγχοντος τα δημόσια έγγραφα. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης, έχουμε περιπτώσεις ένδικων διαφορών για κάποια έγγραφα τα οποία δεν πέρασαν από τον δέοντα έλεγχο. Έφεραν ευθύνες επομένως οι αρμόδιες αρχές. Δεν είναι δυνατόν να υπεκφύγουν αυτές τις ευθύνης με οποιοδήποτε σύστημα. Γιατί ακριβώς ε, το ότι κάποιο είναι αμελής δυνατόν να έχουμε συνέπειε ε, αστικού αλλά και ποινικού δικαίου. Τώρα, αυτό που προαναφέρατε πρόεδρε για την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ. Δεν μπορώ να επεκταθώ στο ποιοι είναι οι δεσμοί που κρατούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη. Αλλά πάντως θα πρέπει να πούμε ότι η κάθε εθνική ενωμή τάξη περιφρουρεί τη δική της προσέγγιση στο δίκαιο. Και αυτό είναι θεμητό. Να, ε, αναφέρθηκε προηγουμένως η προοπτική της κωδικοποίησης. αν υπήρχε μια κωδικοποίηση, μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση, αυτό θα έφερνε μια επανάσταση στην προσέγγιση του ιδιωτικού διεθνέ δικαίου. Όλοι θα συμφωνούσαν για έναν τέτοιο κώδικα, μια τέτοια κωδικοποίηση. Ίσως στο μέλλον επερχόμενες γενναίες το καταφέρουν. Αν εδώ μιλούμε για την τύχη των εγγράφων των σχετικών με την οικογενική κατάσταση, τότε μας ε, καθοδηγεί το άρθρο 21 που δίνει μια τριετία όσον αφορά τη διαπίστωση της ε, κατάστασης του καθεστώτος της γνησιότητάς του. Έτσι κανείς θα πρέπει να ερμηνεύσει τον κανονισμό. γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ζωή των Ευρωπαίων ευκολότερη. Άρα αξίζει να το προσπαθήσουμε. Α, πάρα πολύ σοφά λόγια, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτή μας η συζήτηση, αυτή η φάση των εισηγήσεων. Σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Πρόεδρε, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε για ένα καφεδάκι, ένα μικρό διάλειμμα. Άλλωστε πρόκειται περί συνταγματικού δικαιώματος. και 11 και 20 ξαναρχίζουμε. Έξω από την αίθουσα υπάρχει καφεδάκι. What time is it to say? It's 8? Oh, well, nice. That's okay, yeah.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 ενδιαφέρονται, παρακαλέσια, για τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που θα εξετάσουμε τώρα, παρακαλούνται να καθίσουν. Σας ε, ευχαριστώ. Καλωσορίζω την κυρία, ε, την κυρία Βέντερχόστ από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ε, διότι ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της ε, δυνατότητας ενός ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου. Ποιος είναι ο στόχος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στον 21ο αιώνα πολίτες που κυκλοφορούν ελεύθερα, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, πεθαίνουν εκτός ε, της χώρας όπου γεννήθηκαν. 13% ε, των νέων γάμων έχουν μια τέτοια διεθνή διάσταση και το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο για τις καταχωρισμένες εταιρικέ ε, σχέσεις. Το κόστος ε, που συνδέεται με τα, τη διευθέτηση των διαφορών ε, των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων ανέρχεται σε 1,1 δις το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εσωτερική αγορά στο βαθμό που είναι μια, ένας ενιαίος χώρος ελευθερίας, ε, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Κοιτάξτε το χάρτη. Είναι η κατάσταση όπως έχει σήμερα παρότι η κατάσταση δεν είναι πάντοτε περίπλοκη, τα διεθνή ζευγάρια, στα αποφύσουμε έτσι, καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία προβλήματα. Πρώτον, ε, οι σύζυγοι που βρίσκονται προεκπλήξεως ε, όταν βρεθούν σε μία άλλη χώρα. Το, ο συνήθις τόπος διαμονής καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό, αν ναι, σημειωθεί αλλαγή στο συνήθι τόπο διαμονής αυτόματα, αλλάζει και το εφαρμοστέο δίκαιο. Βάζει του κανονισμού Ρώμη 3, παραδείγματος χαρή, αν μετακομίσει κάποιος σε άλλο κράτος μέλος, ε, ο κρίνεται ένα διαφορετικό γαμικό καθεστώς και καταλαβαίνετε πόσο έκπληκτη είναι η σύζυγη, ε, ένα αυστριακό ζευγάρι παραδείγματο χάρη που μετακομίζει στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το δίκαιο για τα διαζύγια ανάμεσα στις δύο χώρες και όπως βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα στη διαφάνεια μπορεί αυτό να επιφυλάξει πολύ μεγάλες εκπλήξεις για το ζευγάρι και κυρίως για το πιο αδύναμο ε, μέρος. Ας φανταστούμε ότι στην χώρα προέλευσης ε, το κληρονομικό δίκαιο ε, αναγνωρίζει δικαιώματα σε κάποιον που συζεί έναν εταίρο που συζεί αλλά δεν έχει ε, παντρευτεί και στη συνέχεια μετακομίσει τον λόγο άτομο σε μια χώρα όπου δεν αναγνωρίζονται τέτοια δικαιώματα γίνεται εφαρμοστέο το δίκαιο της χώρας διαμονής, συνήθως διαμονής ε, ε, και χάνονται όλα τα δικαιώματα. Ας περάσουμε τώρα στο φόρουμ shopping. Αυτά σχετίζονται με τα προβλήματα του κανονισμού Ρώμη 2α. Μπορεί να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για έναν από τους εταίρους ή συζύγους να κινήσει τη διαδικασία ταχύτατα σε ένα φόρουμ που διαφυλάτει εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Όταν έχετε προγαμίο σύμφωνο, παραδείγματο χάρη, αυτό είναι ισχυρό κίνητρο να σπεύσει ε, ένα από τα δύο μέρη και να κινήσει τη διαδικασία σε μια χώρα όπου τέτοια προγαμία σύμφωνα δεν κρίνονται απολύτως δεσμευτικά. Το τρίτο πρόβλημα, και αυτό ίσως είναι και το σοβαρότερο, είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα στα εφαρμοστέα δίκαια και τα φόρα. Δηλαδή, ακόμη και σε διασυνοριακές περιπτώσεις ε, μπορεί να έχουμε διάφορα φορά με δύο-τρία διαφορετικά εφαρμοστέα δίκαια. Θα ήθελα να πάρω ένα παράδειγμα ενός ζευγαριού παντρεύτηκε στη Γερμανία και συνέχεια μετακόμισε στην Αυστρία, παίρνει διαζύγιο και ε, ο σύζυγος παραδείγματος χάρη μετακομίζει στην Ολλανδία και ξεκινάει εκεί τη διαδικασία διαζύγιο. Δεν είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Έχουμε τις, τα περιουσιακά στοιχεία, έχουμε σπίτι, κοινό, ένα παιδί στο γάμο και χωρίς να μπω μέσα σε λεπτομέρειες, ε, είναι περίτω, ε, υπάρχει Υπάρχουν διάφορα φορά και διάφορα εφαρμοστέα δίκαια, το γερμανικό, το αυστριακό και το ολλανδικό, με πάρα πολλά ερωτηματικά, διότι δεν έχουν ρυθμιστεί όλα και υπάρχουν σοβαρές ανακολουθίες. Ε, σύγκρουση δικαίων, λοιπόν. Τελικά έχουν βρεθεί εξαιρετικά περίπλοκες λύσεις για αυτές τις περιπτώσεις, όμως τα δικαστικά έξοδα ε, είναι εξαιρετικά υψηλά και είναι ε, πάρα πολύ χρονοβόρη η διαδικασία. Δεν συνάδει αυτό με τις πρακτικές του 21ου αιώνα. Ε, λοιπόν, ε, δεν μπορεί να αποτελεί αυτό εμπόδιο για κάποιον που θέλει να μετακομίσει και να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και να μην γνωρίζει τις νομικές συνέπειες ε, των πράξεών του. Ποια θα ήταν η λύση για αυτό το πρόβλημα. Ε, μια τομεακή κωδικοποίηση της σύγκρουσης δικαίων ο καθηγητής Φανχάη αναφέρθηκε σε αυτό, ή ε, ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γάμο, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, τουλάχιστον ε, στο εγγύσμα. Μία άλλη ιδέα θα ήταν να ενισχύσουμε την αυτονομία των μερών, δηλαδή να κινηθούμε προς μεγαλύτερη αυτονομία. Όταν εξετάζουμε τα υφιστάμενα εργαλεία και συγκεκριμένα ε, στον κανονισμό για τις περιουσιακές σχέσεις ε, των συζύγων ε, και αν αναθεωρηθεί ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α θα μπορούν να επιλέγουν εκ των προτέρων τα μέρη, το εφαρμοστέο δίκαιο, αποφεύγοντας έτσι τις εξαιρετικά δυσμενικές ασθενείς επιπτώσεις που μόλις διαπιστώσαμε. Επιλογή του δικαστηρίου λοιπόν και του εφαρμοστείου δικαίου. Να, αυτό θα μπορούσε να είναι ε, μία λύση και ε, σε σχέση με τα ε, πρόγραμμια σύμφωνα θα μπορούσε αυτό να αποδειχθεί μια ικανοποιητική λύση. Λοιπόν, αν υπάρχει αυτή η λύση, γιατί δεν τη χρησιμοποιούν τα ζευγάρια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, δεν γνωρίζουν αυτέ τι ανελεκτικέ λύσει. Δεν ε, ε, συνειδητοποιούν ότι είναι στη διάθεσή τους αυτές ε, οι νομικέ λύσει. Στη συνέχεια μπορεί να δημιουργήσει αυτό πρόβλημα στη σχέση. Επίση, δεν ξέρετε αν θα είναι σε προσιτή τιμή η δικαστική συνδρομή για να κατανοήσετε όλες αυτές τις διαφορετικές λύσεις. Προτείνω λοιπόν να έχουμε ευρωπαϊκές πρότυπες διατάξεις ε, για την επιλογή του δικαστηρίου και του εφαρμοστέου δικαίου και... Αυτό θα είναι προαιρετικό. Ε, να προβλέπεται η οικογενειακή διαμεσολάβηση θα πρέπει να συνειδητοποιούν τα μέρη κάθε φορά που συνάπτεται ένας γάμος ε, ή καταχωρίζεται μια εταιρική σχέση ή ε, μια διασυνοριακή αλλαγή ε, του συνήθου τόπου διαμονής ή καταγραφή μιας γέννηση, τότε θα προβλέπετε ένα μονοαπευθυντικό πακέτο διασυνοριακό που θα οδηγεί σε εφαρμογή ενός ενιαίου δικαίου. Ένα δεύτερο βήμα θα ήταν ενδεχομένως πρότυπες συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ζητήματα ουσιαστικού και οικογενειακού δικαίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο και ενδεχομένως θα αποβεί περισσότερο προβληματικό. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι σε συνεργασία με την καθηγήτρια Κατερίνα Ουλαμβέρκη, που είναι καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής για το Οικογενειακό Δίκαιο, συντάξαμε αυτό την πρόταση και θα μπορούσε να λειτουργήσει υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή We thank you, Professor. Εμείς ευχαριστούμε, καθηγητά, λέει Και τώρα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Κουρτ Λέχνερ Ποιο είναι εισηγητής για τον κανονισμό για τις διαθήκες αλλά επίσης έχουμε εδώ και την κυρία ε, Εύ Πούτερ που είναι νομική σύμβουλος του Συλλόγου Συμβολιογράφων της Εστονίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Μέχρι πριν από τρία χρόνια ήμουν εδώ ως βουλευτής, ευρωβουλευτής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το έργο το οποίο έχουμε μπροστά μας και, και εγώ ο ίδιος συνέβαλα σε αυτό το έργο. Μετά από κάποια απόσταση που πήρα μπορώ να κάνω και κάποια κριτική. Έχω και εγώ κάποιες διαφάνειες. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω τον κανονισμό, γιατί εδώ και τρία χρόνια ισχύει. Εφαρμόζεται και από τις 17 ε, Αυγούστου. Ελπίζω να μην μας αγγίξει εμάς άμεσα όλους. Θα υπάρχουν και στο μέλλον προβλήματα. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα στην παρούσα φάση. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Βέντε Χόρστ ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ε, πλήττεται και ο ένας από τους δύο συντρόφους εφόσον δεν έχουν, δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα αυτά. Αυτό φυσικά οδηγεί σε προβλήματα. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποια στοιχεία. για τον κανονισμό. Πρόκειται για ένα συνδυασμό της τελευταίας διάμονης και της ελεύθερης ε, επιλογής ε, δικαιοδοσίας. Αυτό είναι το θέμα του κανονισμού. Η βιβλιογραφία είναι τεράστια. τότε τα πρώτα σχόλια, μας ε, προκαλεί εντύπωση πόσο μεγάλο είναι το εύρος των προβλημάτων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για τον κανονικό πολίτη ο κανονισμός θα πρέπει να είναι κατανοητός και εύληπτος. Δεν χρειάζεται να ξέρει οι τεχνικές λεπτομέρειες. Αν ε, το μόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι ότι αν για παράδειγμα χαλάσει ο γάμος μου έχω δικαίωμα να διαλέξω μεταξύ του τόπου διαμονής ή του, της πατρίδας μου σε ό,τι αφορά την ομολογία την ε, δικαιοδοσία. Και καλό είναι επίσης να υπάρχουν όσο πιο λίγες ε, μεμονωμένες νομοθεσίες γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ήταν σημαντικό να μην οριστεί η τελευταία κατοικία, η συνήθις διαμονή. Αυτό ορίζεται και σε... Μάλλον δεν ορίζεται και σε άλλους κανονισμούς και ευρωπαϊκούς αλλά και των κρατών μελών σε νομοθετήματα το θέμα της ε, διαμονής, του τόπου διαμονής. Και νομίζω ότι ο όρος αυτό δεν μπορεί να είναι ενιαίος για όλους. Σε οριακές περιπτώσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον κανονισμό διατροφή, σε ό,τι αφορά τον τόπο διανομής ενό παιδιού. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαφορετική αντιμετώπιση. Κατά τα άλλα θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα πλαίσιο ενός ξεχωριστού EPR, για παράδειγμα. Στην παράγραφο 21, παράγραφος 2 ο συμβιβασμό που πετέχθηκε τελευταία δεν μπορεί να δικαιολογήσει αποκλειστικά την δικαιοδοσία. Σκόπιμα έγινε αυτό. Δηλαδή το αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό του τελευταίου τόπου διαμονής. Θα πρέπει να εφαρμόσει σε, περίπτωση, σε κάποιες περιπτώσεις την νομοθεσία μιας άλλης χώρας. Ο Αντιπρόεδρος ανέφερε το θέμα της υπηκορητικότητας, γιατί το κληρονομικό δίκαιο ουσιαστικά είναι ένα θέμα κουλτούρας των κρατών μελών και ο κανονισμός προσπαθεί να ε, περιορίσει τις παρεμβάσεις όσο πιο περισμένες γίνεται, γιατί οι συγκρούσεις ε, έμεσα επηρεάζουν το κληρονομικό δίκαιο και μπορεί να προκαλέσουν και σύγκληση το σημαντικό είναι να μην πληχθεί καμία νομοθεσία και να υπάρξουν τα εργαλεία που υπήρχαν έως τώρα. Ο κύριος Λαγκάρτ είπε ότι ο κανονισμός είναι μια πραγματική επανάσταση και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι καινούριο για όλους. Επειδή ήταν επιτυχής επειδή επικεντρωθήκαμε στα καινούργια στοιχεία. Δεν, προσπαθήκαμε, δεν προσπαθήσαμε να εξαγάγουμε τα παλιά στοιχεία ο καθένας από τη χώρα του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη σύνθεση του κανονισμού. προκειμένου να υπάρχει καλή συνεργασία των διατάξεων. Μπορεί να είναι ενδιαφέρουσε οι εθνικές προβλέψεις, αλλά δεν έχουν εφαρμογή εδώ. Επειδή μιλάμε για πολίτες, να υποδείξω και το φορολογικό ζήτημα. Φυσικά ο κανονισμός δεν μπορεί να ορίσει φορολογικές διατάξεις, αλλά ο κόσμος το ζει αυτό στο πεζί του και εμέσως ε, ε, επηρεάζει τα θέματα αυτά, γιατί φυσικά έχει να κάνει με την ε, διάθεση της κληρονομιάς, των περιουσιακών στοιχείων και δυστυχώς θεωρώ ότι στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει προθυμία να πάμε σε επίπεδο ε, οδηγίας πλαισίου. Και επίσης επικριτικά να αναφέρω ότι στα κράτη-μέλη δεν έχουν διοργανωθεί ενημερωτικές εκστρατείες που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει συμβεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντά της και πολλοί δικηγόροι, συμβολιογράφοι κάνουν ε, καταρτήσεις, εκπαιδεύσεις, ε, μετεκπαιδεύσεις, αλλά το λέω αυτό προς τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια ότι πρέπει να κάνουν κάτι και τα Εθνικά Κοινοβούλια για να ενημερώσουν τους πολίτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Δανία δεν συμμετέχουν στην ε, κανονισμό. Κρίμα. Και ο κανονισμός ο ίδιος δεν ορίζει ξεκάθαρα και ρητά ότι πρόκειται για τρίτες χώρες. Σε άλλους κανονισμούς προβλέπεται και αναφέρεται ρητά αυτό. Ποιο είναι το συμπέρασμα λοιπόν αν άλλοι κανονισμοί και άλλα νομοθετήματα ρητά αναφέρουν αυτέ τι χώρε ω τρίτε χώρε ενώ δεν αναφέρεται αυτό στο συγκεκριμένο κράτο, τα συγκεκριμένα κράτη. Ε, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο και να πω ότι ο τόπο δεν είναι ίδιο με τον τόπο κατοικία, όπω ε, στις ε, είπα και αυτό ενδεχομένω να προκαλέσει μεγάλε συγκρούσει. Ένα σημαντικό ζήτημα που μας ξεφεύγει είναι το θέμα των κρατικών ε, συνθήκων, σε πόσο και πόσο συγκρούονται με τρίτες χώρες. Αυτό αναφέρεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας του 3150. Αυτό οδηγεί σε μαζικά προβλήματα. Δεν έχω χρόνο να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Οι εθνικές νομοθεσίες εκτελούνται από τα εθνικά δικαστήρια ανεξαρτήτως των συνθήκων. Και καλό θα ήταν να είναι ερμηνεύονται και να τηρούνται περιοριστικά αυτές οι εθνομοθετικές νομοθεσίες. Ακόμα καλύτερο ασφαλώς ότι θα ήταν να καταργηθούν. Από πολιτική άποψη είναι σωστό ασφαλώ αν τα κράτη και το ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό από κοινού. Για τη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει διμερή σύμβαση με την Τουρκία, η Ιταλία επίση, τα πρώην κράτη της Σοβιτικής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε να τα επεξεργαστούμε. Και το λέω αυτό και σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά. Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να πω μια τελευταία κουβέντα. Εγώ φοβάμαι ε, ότι είναι πολύ ευρύ το θέμα, όπως και φοβόμασταν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε τα, στα αξιώματα, στα αιτήματα των εθνικών αντιπροσωπιών. Και αυτό το έχω δει και σε τη προστασία του καταναλωτή. Ο καθένα τι θέλει να τεθεί το δικό του το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση να απαντηθεί το δικό του το πρόβλημα. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι όλα αυτά προστίθονται το ένα στο άλλο και το αποτέλεσμα δεν είναι εύληπτο. Θα δούμε. Θα δούμε πώς ε, θα δημορφωθεί αυτό στο μέλλον και κατά πόσον σε συνεργασία, σε, σε, συνάρτηση και με άλλα νομικά προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει το δικαστήριο θα επικρατήσει αυτό το ευρωπαϊκό έντυπο. Υπάρχουν και μερικές συγκρούσεις ε, σε ό,τι αφορά τη στοχοθέτηση. Κάποιες εξ αυτών θεωρώ ότι με διαπραγματεύσεις μπορούν να επιληθούν. Να υπάρξουν διευκρινήσεις, να περιμένουμε καταρχάς λίγο να γίνουν κάποιες πρακτικές αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά. Εγώ θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δικαίωμα του κληρονόμου για την επιλογή του δικαίου. Και αυτό που θα ήταν κατεπήγον να ολοκληρωθεί και ο κανονισμός για τα δικαιώματα αγαθών, γιατί υπάρχουν πολλές ε, συναρτήσεις με την, ε, τον κανονισμό για τις ε, κληρονομιές. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει... Κύριε Πόντρο, σας ευχαριστώ που μου την ευκαιρία να παρίσταμε εδώ. Πριν σας μιλήσω για τις διαθήκες, πρέπει να σας πω ότι έχω εργαστεί και στα πλαίσια του Σουλευρικού Συλλόγου. Και οπότε έχω ασχοληθεί και με το θέμα της ε, επικύρωσης και πίστος γνησιότητας των διαθήκων. Στην Εστονία, εδώ και χρόνια, οι διαθήκες περιθυμίζονται ανάλογα με την τελευταία κατοικία. Και το εφαρμοστείο δίκαιο είναι το δίκαιο της ε, χώρας τελευταίας κατοικίας του αποθανόντος. Να σας πω ποια είναι η εμπειρία μας όσον αφορά επομένως τον κανονισμό και ό,τι καλύπτει εξαρτάται ε, από την ηθαγένεια του θανόντος και από το που βρίσκονται τα ε, ακίνητα που καλύπτονται από την Διαθήκη. Θα είναι ευκολότερο για τους κληρονόμους τώρα. Δεν θα χρειάζεται πια να γίνονται κάποιες δίκες σε διαφορετικά κράτη-μέλη και άλλες διαδικαστικές ενέργειες. Επίσης, αυτός ο κανονισμός θεσπίζει συγκεκριμένου κανόνες για την διαπίστωση γνησιότητα τη διαθήκη. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όποτε κανείς συντάσσει Διαθήκη. Τώρα, για το εφαρμοστείο δίκαιο για την δοσηδικία κριτήριο θα είναι η τελευταία κατοικία του θανόντος. Η δυσκολία βέβαια είναι ότι ο κανονισμός δεν ξεκαθαρίζει τι είναι συνήθις τόπος διαμονής ή ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί ποιος τόπος είναι αυτή η διαμονή. έχει κρίνει από αυτού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι υπάρχει συγκεκριμένη έννοια διαμονής που πρέπει να χρησιμοποιείται για το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορεί κανείς να έχει συνήθει διαμονή σε περισσότερα από ένα κρατημέλιο. Για ακίνητα, για πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων κλπ. Όλα αυτά είναι στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, ούτω ώστε να καθοριστεί ο τόπος συνήθους διαμονής κάποιου. Η πρόθεση μονίμου κατοικίας επίσης λαμβάνεται υπόψη αν κρατήσει κάποια χρόνια. Και να κρίνουμε τώρα κατά πόσον ο Θανόν είχε σύνθη ε, διαμονή θα πρέπει ε, ε, σε κάποιο κράτος μέλος θα πρέπει να τον υπόψη κάποια κριτήρια, τα 11 κριτήρια που προβλέπονται. Τώρα οι ωφελούμενοι από την κληρονομιά και από την Διαθήκη αυτοί έχουν το άνομο συμφέρον να καθορίσουν ποια είναι η συνηθής διαμονή. Πάντως, ε, αποδεικτικό στοιχείο δεν θεωρείται πιστοποιητικό γέννησης. Στη χώρα μας έχει κρυφεί ότι η πρόθεση των διαδίκων θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Έχουμε τώρα κάποιες διασυνοριακές περιπτώσεις. Οπότε, οι κληρονόμοι ισχυρίζονται ότι ο Θανόν είχε περισσότερες, περισσότερους τόπους διαμονής. Πάντως, εμείς πάντοτε προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα στο να ε, ξεκαθαριστεί η υπόθεση στην Εστονία, γιατί θα ήταν τα πράγματα πιο περίπλοκα και πιο ακριβά, εάν ε, η δίκη γινόταν σε άλλο ε, κράτος μέλος. Θα υπήρχε και θέμα φόρου κληρονομίας. Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό της ε, Διαθήκης, όπως το ορίζει ο κανονισμός, μπορεί να αποτελέσει απόδειξη για το ότι έχουν ε, γίνει οι διαδικασίες και το ότι οι δικαιούχοι της ε, Διαθήκης τελικά έχουν καθοριστεί το ποιοι είναι. Πάντως, έτσι δεν έχουμε δημιουργία κάποιων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αποδείξουν αυτοί οι δικαιούχοι ότι έκαναν ό,τι απαιτείται και με αυτές τις διαδικασίες προέταξαν την αξίωσή τους σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος. Έχουν επίσης την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχουν. Και ιδίω στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία σε άλλη χώρα μέλος. Μετά από χρόνια που έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη διαδικασία, τότε ακόμα, ακόμα για να έχουμε αίτηση για επιστοποιητικό σύμφωνα με τον κανονισμό. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι διαδικασίες. Εθνικό ή ευρωπαϊκό τέτοιο επιστοποιητικό, ανεξάρτητα του αν έχουν γίνει διαδικασίες δικαστικά ή εξοδικαστικά. θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμό όσον αφορά τη δόση δικαία και όσον αφορά το φαρμαστείο δίκαιο. Οπότε και έχουμε με τότε την έκδοση του πιστοποιητικού. Υπάρχει εδώ μια σειρά υποχρεώσεων που συντρέχουν και όλα αυτά ισχύουν μόνο στην περίπτωση που οι εθνικέ αρχέ έχουν ε, πρόθεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για τα ζητήματα του κανονισμού. Θα αρχίσει η διαδικασία λοιπόν από το αρμόδιο δικαστήριο για να βεβαιωθούμε το ότι το δικαστήριο της Γενικής Δοσηδικίας δεν έχει αρχίσει παράλληλα διαδικασίες, θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της εύλογης αμφιβολίας. Και έτσι το δικαστήριο στο οποίο έχουν προσφύγει ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαπιστώσει το τι γίνεται με το δικαστήριο Γενικής Δοσηδικίας Στην Εστονία Ας πούμε, έχουμε κάποιους από την Φιλανδία οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το δικαστήριο, το αρμόδιο. Και αυτό που λαμβάνει την υπόψη είναι ποια ήταν η τελευταία διαμονή του θανόντος. Και πριν εκδοθεί το πιστοποιητικό, θα πρέπει να γίνει έρευνα από τις αρχές για το κατά πόσον υπάρχει διαθήκη σε άλλο κράτος μέλος. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι σύμφωνα με τον κανονισμό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητούν από άλλο κράτος μέλος πληροφορίες αλλά μόνο όσον αφορά τα του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού. Ο δε κανονισμός δεν προβλέπει υποχρέωση παροχής πληροφοριών όταν αυτό απαγορεύεται από το εθνικό δίκαιο. Άρα, σε κάποιες επιπτώσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν οι διαδικασίες και από την άλλη μεριά οι δικαιούχοι θα πρέπει να ταξιδέψουν σε άλλο κράτος μέλος τόσο ώστε να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους που παρέχονται σε άλλη διαθήκη. Ε, τώρα σε που υπάρχει νεότερη διαθήκη θα πρέπει να αναζητηθεί τώρα ε, το ποιο είναι υπεύθυνο για το ότι δεν αναζητηθεί η νεότερη διαθήκη. Φταίνε οι αρχέ ή φταίνε οι κληρονόμοι. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος και το ότι το εφαρμοστείο δίκαιο θα επιλέγεται με τα ίδια κριτήρια και παντού. Λιγότερη γραφειοκρατία χρειάζεται. Για τις επικυρώσεις, για την αναγνώριση των αλλοδαπών αποφάσεων και για το πιστοποιητικό. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση. Από την άλλη μεριά βέβαια, ακριβώς όπως ε, οι αναλύσεις έχουν καταδείξει, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα ε, για το ότι οι αρχές οι οποίες πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις διαθήκες ε, θα τα αντιμετωπίσουν για την εφαρμογή του κανονισμού. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές ποιοι δικαιούνται να συμπήξουν μια συμφωνία επιλογής διαστηρίου και όσον αφορά την μεταφορά αρμοδιότητας και ποιος επίσης μπορεί να ενίσταται ε, άλλοι άλλη σε άλλο κράτος μέλος, κάποιοι πιστωτές του θανόντος. Δεν προκύπτουν αυτά από τον κανονισμό. Επομένως, έχει κάποια παραθυράκια, έχει κάποια ερωτηματικά αναπάντητα ε, ο κανονισμός. Όλα αυτά θα πρέπει να επιληθούν είτε με νομολογία είτε με άλλο καινούργιο κανονισμό. Thank you very much for your... Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Ρωτώ απλώς ε, Έχετε ερωτήσεις για τους διακεκριμένους ομιλητές μας, ε, είτε ε, οι βουλευτές ή κάποιος άλλος. Φαίνεται ότι ήταν πληρέστατες ε, οι παρουσιάσεις. Εσείς θα θέσετε ερώτημα στον εαυτό σας. Όχι, Πρόεδρε. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να επανέλθω για, σε ένα θέμα και για τις εργασίες της Επιτροπής εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα θέμα το οποίο δεν ανέφερα λόγω χρονικών περιορισμών. Συνολικά, θεωρείται βασικό μειονέκτημα του κανονισμού το εξή ότι η επιλογή, τόπου, η επιλογή δικαίου περιορίζεται μόνο στην ηθαγένεια. Και ο λόγος είναι ότι δεν επιτρεπόταν η επιλογή του δικαίου για τον τόπο συνήθω διαμονή. Δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου τότε. Θεωρώ ότι όταν έχουν συνηθίσει πλέον τα κράτη-μέλη στην ε, τρέχουσα κατάσταση, καλό θα ήταν να υπάρχει η, επιλογή, η δυνατότητα επιλογή του δικαίου του τόπου συνήθω διαμονή. Υπό στενή έννοια. Δέκα χρόνια δηλαδή τουλάχιστον διαμονή και κυρίως όταν πρόκειται σε, για γάμους ε, διπλής υπηκότητας. Να μπορεί να επιτρέψει δηλαδή ο ένας από τους δύο να επιλεχθεί το δίκαιο του άλλου. Στην αρχή λοιπόν ήταν πολύ μεγάλες οι ανησυχίες, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη μελλοντική μεταξύλιξη του κανονισμού. Και αντίθετα με αυτά που είπε η συνάδελφος Πίτερ, σημαντικό είναι σε θέμα αρμοδιοτήτων αν ε, υπάρχει επιλογή του, της δικαιοδοκησίας να ορίσουμε ένα στενό κύκλο συμμετεχόντων. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να δώσουμε το δικαίωμα στους κληρονόμους αν υπάρχει επιλογή του δικαίου να ορίσουν αυτοί και τη δικαιοδοσία τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα θα τα λύναμε. Σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να προσθέσω αυτά τα στοιχεία. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Mrs. Potter, please. Thank you. I would like... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Τα άτομα έχουν δικαίωμα να ορίσουν τη διαθήκη τους και να επιλέξουν την ε, ότι το δίκαιο του, της χώρας της οποίας τις υπηκότητας έχουν να ισχύσει για τη διαθήκη τους. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι όταν γίνεται η επιλογή αυτή, γιατί όταν κάποιο καταρτίζει τη διαθήκη του και έχει δυνατότητα να διαλέξει μεταξύ διαφορετικών δικαίων, προφανώ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο του εκάστοτε δικαίου στην κληρονομιά. Γιατί αν η διαθήκη, για παράδειγμα, καταρτιστεί στην Εστονία, αλλά το άτομο ζει τη στιγμή του θανάτου στην Ολλανδία, η τελευταία διαθήκη θα καταρτιστεί σύμφωνα με τους νόμους της Εστονίας, αλλά όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία κληροδότησης θα γίνει ερμηνεία σύμφωνα με το Ολλανδικό Δίκαιο. Αυτό λοιπόν θα περιπλέξει την κατάσταση και στην τελική ανάλυση τι θα συμβεί. Οι τελικές επιθυμίες του αποθανόντος δεν θα γίνουν σεβαστές. Και επίση, ένα άλλο κίνδυνο που ενέχεται στον κανονισμό επιτρέπει στα άτομα να επιλέξουν την εθνικότητα, την υπηκότητα που έχουν τη στιγμή του θανάτου. Αυτό τι σημαίνει η υπηκότητα που θα υιοθετηθεί στο μέλλον. Είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς πώς θα ερμηνευθεί σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του άγνωστου κράτους σε ό,τι αφορά την Διαθήκη. Άρα ίσως αυτό καλό θα ήταν να το... Μην το συστήνουμε στους πελάτες μας στην κατάρτιση των διαθήκων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σκλάνση. Thank you. Um, of course... Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει προσυπογράψει αυτό το σχέδιο οργανισμού. Οπότε πέρα μάλλον παρήσακτος είμαι εγώ. Αλλά, α, σκεπτόμουν αυτά τα οποία μας είπατε πριν για το θέμα της ε, ηθαγένειας, της ε, διαμονής και εάν προσχωρούσε το Ηνωμένο Βασίλειο τότε θα υπήρχε πρόβλημα γιατί πρόκειται για κράτος με πολλές δοσιδικίες και στο κληρονομικό δίκαιο. Βέβαια, όπως είπαμε, το βασικό κριτήριο είναι η κατοικία του θανόντος. Και έχουμε πλούσια νομολογία από αυτού. Και όταν λέω για κατοικία, ενώ το που είναι η νόμιμη κατοικία του θανόντος. Έτσι καθορίζεται η δοσηδικία. Αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει τον απλό κόσμο, αλλά τέλος πάντων θα έπρεπε να δούμε πώς αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Yes, madam. Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, κυρία Πέτρου που αναφέρθηκε σε αυτά τα επιπρόσθετα σημεία, διότι όντως ε, ορισμένε φορές έχουμε τεράστια προβλήματα, διότι ε, ένα Ολλανδικό δικαστήριο θα ερμηνεύσει το ιστονικό δίκαιο, όπως σωστά είπατε, και ένα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε με τις ευρωπαϊκές πρότυπες διατάξεις. Θα υπάρχει επιλογή δικαίου για τα κληρονομικά ζητήματα μεταξύ άλλων και έτσι δεν θα υπάρχουν αυτές οι διαφορές που σωστά υποδείξατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή μας πρωινή σύσκεψη στις 2.30 θα επιστρέψουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6 ακριβώς και άρα θα είμαστε πιεσμένοι ως προς το πρόγραμμα. Παρακαλώ να αρχίσουμε ακριβώς την ώρα μας. Οι εμπειρογνώμονες που θέλουν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλύματος να φύγουν από το κτίριο έχουν φυσικά τη δυνατότητα, όμως ε, θα πρέπει... Θα πρέπει να συναντηθείτε με το προσωπικό από τις 2 μέχρι τις 2.30 για να ε, σας βγάλουμε την κάρτα σας και να μπορείτε να ξαναμπείτε στο κτίριο. Αλλιώς ε, δεν θα είναι δυνατόν διότι υπάρχει ένα αυξημένο σύστημα, ενισχυμένο σύστημα ασφαλείας. Ε, ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στις 2.30.